Καλησπέρα όλοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω είναι και πέντε. Απογευματινή συνεδρία τη Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα έχουμε την έγκριση του σχεδίου ημερήσια διάταξη που είναι στα αγγλικά. Διαβιβάστηκε στι 20 Οκτωβρίου του 2009 και μπορείτε να το βρείτε στου φακέλου σα. Δημοσιεύτηκε και στην ισοσελίδα μας. Έχουμε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης των προηγούμενων συνεδριάσεων 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Διαβιβάστησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούνται ως εγκεκριμένα και τα πρακτικά. Στο σημείο 3 έχουμε web streaming, έχετε τις γλώσσε, έχουμε ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας για αύριο. Θυμηθείτε να έχετε, διότι αύριο θα γίνει η ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο και επιθυμίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα, 10 Νοεμβρίου του 2009, θα γίνει η παρουσίαση της ετήσιας εκθέσεως του ελεκτικού συνεδρίου. Σας λέγω ότι 22 Οκτωβρίου του 2009 ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών του Ολλανδικού Κοινοβουλίου των Κάτω Χωρών έστειλε μια επιστολή για να συμμετάσχουμε σε μια διάσκεψη σημαντική κατά την απόψή μου για τη βελτίωση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι οργανωτέ της διασκέψη αυτή θέλουν να αφοστείλουν πρόσκληση και στου αντιπροέδρου της Επιτροπής. Εάν οι τέσσερι αντιπρόεδροι δεν είναι διαθέσιμοι ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν, οι οργανωτέ δέχονται τη συμμετοχή άλλων μελών της επιτροπή. Έχουμε προθεσμία μέχρι το Δεκέμβριο, όποιος ενδιαφέρεται ή οι αντιπρόεδροι ή κάποιοι από τα μέλη της Επιτροπής ας ειδοποιήσουν σχετικά την γραμματεία για να συμμετάσχουν. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας θα ήθελα να χαιρετήσω τρία νέα μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής, δύο νέους βοηθούς, την κυρία Σιλβάνα Τζάμιτ και την κυρία Ροζαμαρή Ελφκουίστ και την κυρία Έλενα Μαϊνάρντι, μέλο τη διοίκηση, και στου τρει απευθύνω τον πιο θερμό μου χαιρετισμό και εύχομαι καλή δουλειά σε μια σημαντική επιτροπή που είναι η δική μα. Στο τέταρτο σημείο τη ημερήσια διάταξη, Βλέπουμε το θέμα μας που αφορά την απαλλαγή του οικονομικού έτους 2007. Θα ζητούσα από τον εισηγητή, τον κύριο Αοντή, αν θέλει να μιλήσει πρώτος ή να μιλήσει πρώτος ο Επίτροπος, ο κύριος Κάλλας. Λοιπόν, ο Επίτροπος ο κύριος Κάλλας ε, μπορεί να πάρει το λόγο, το χαιρετίζω, καλώς ήρθατε και παρακαλώ να προβείτε στην παρουσίασή σας. Έχετε το λόγο κύριε Κάλλας. Thank you much, Mr. Ευχαριστώ αξιότιμοι ευρωβουλευτές αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία συμφωνία Καταρχήν ότι θα παρουσιάσω όλες μου τις παρατηρήσεις από την αρχή, δηλαδή θα ξεκινήσω με το σχέδιο ψηφίσματος και μετά θα προχωρήσω στην παρουσίαση της έκθεσης. Ε, συμφωνείτε? Καλά έχω καταλάβει. Ωραία. Οπότε θα προσπαθήσω να καλύψω και τα δύο θέματα. Για το, ψήφισμα για την απαλλογή του 2007 έχει πάνω από 200 παραγράφους και αιτήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δέχεται αρκεί ε, να μην αντιτίθενται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και όλα αυτά συνάδουν με την ανακοίνωση της 28ης Οκτωβρίου. Θα αναφερθώ εδώ σε δύο θέματα. Καταρχάς την ουσία του, ε, της περίληψης η οποία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ε, και ε, ε κατά πολύ τα κράτη-μέλη μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διότι μέχρι στιγμής ε, οι περιλήψεις έχουν καταρτιστεί περιμένουμε ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις και θα υπάρξει μία ενημέρωση για την απαλλαγή 2009. Διάφορα κράτη, η, ε, Ουγγαρία, η ε, Κύπρος, η Σλοβακία και άλλες έχουν δεχθεί την πρόταση να έχουν μία εξασφάλιση της αποδόσεως εις ε, την παρουσίαση των στοιχείων και ε, ε, η Ολλανδία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και μία ακόμη χώρα συμπληρώνουν τον κατάλογο των κρατών οι οποίες παρουσιάζουν ένα πιστοποιητικό ακριβία των λογαριασμών τους που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι θα συζητήσετε ε, την εξωτερική έκθεση ε, για τις αξίες εφέτος και πρέπει να σας πω ότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη βελτίωση και θεωρούμε ότι χρειάζεται μία πιο ισχυρή ε, βάση νομική κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ε, τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία από τις 28 Δεκάτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει το, την τελική έκθεση για να ενισχύσει τον υποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες προχωρούν ε, με ε, διάφορες διαδικασίες διορθώσεως είναι θέματα τα οποία θα συζητήσετε με τους αρμόδιους ε, επιτρόπους κατά τη διαδικασία της απαλλαγής οπότε εγώ δεν θα επεκταθώ σε αυτά ε, και τέλος ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα των εσωτερικών λογαριασμών σύμφωνα με ε, το δημοσιονομικό κανονισμό και ε, δεν θα πρέπει ε, να σταματήσουμε να επαγρυπνούμε υπάρχουν ε, οι ε, εκθέσεις τις οποίες έχουν ε, καταρτήσει οι αποδέκτες και έρχομαι τώρα στο θέμα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν διάφορα λάθη και έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να βελτιώσουμε τους λογαριασμούς μας και την την παρουσίασή τους με μέτρα απλοποίησης για τα διαρθρωτικά ταμεία όπως άλλωστε και την δυνατότητα να δηλώνει κανείς ε, ε, τα κόστη με διάφορους τρόπους όπως αποφασίσει το Μάιο του τρέχοντος έτους. Ε, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μία απλοποίηση η οποία θα καταστεί προφανής ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά τις εργασίες της για την τριετή αναθεώρηση ιδίως όσον αφορά τις χορηγήσεις, τους κανόνες επιλεξιμότητος και έχουμε ξεκινήσει μία δημόσια διαβούλευση η οποία είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου και ε, ζητούμε από τους διαχειριστές και τους αποδέκτες των δημοσίων ταμείων να ε, μας σχολιάσουν πώς θα βελτιώσουμε τους κανόνες. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε την νομοθεσία κατά τομέα ε, για να μπορέσει να εφαρμοστεί το 2014 και πιστεύω ότι ε, ο ανεκτός κίνδυνος θα πρέπει να υπερισχύσει κατά τρόπον ώστε να ξέρουμε ποια είναι ε, η ισορροπία στην οποία θα πρέπει να καταλήξει η δημοσιονομική αρχή. Ε, στο θεομέα της ενέργειας των μεταφορών και της βιομηχανίας όπως άλλωστε και της γεωργίας θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία στο δεύτερο εξάμεινο του 2010. Τώρα θέλω να σας παρουσιάσω την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2008 και η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει και πάλι να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και τον εισηγητή κύριο Λιμπεράτσχη. Είναι η τελευταία αυτή παρουσία της ε, τρέχουσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα ε, να χαιρετήσω την ε, δήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει από την αρχή υπεύθυνη για την απαλλαγή να παρουσιάσει το αναγκαίο πιστοποιητικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, απέδειξε ότι είναι δεσμευμένη να συνεχίσει αυτή την εργασία βασιζόμενοι στις ετήσιες εργασίες και εις το πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης εξαρτώμεθα από τις ετήσιες εκθέσεις και το ελεγκτικό συνέδριο μας λέγει ότι οι λογαριασμοί βελτιώνονται κατά τα τελευταία χρόνια χάρη εις την εργασία η οποία έχει γίνει για να βελτιωθεί η παρουσίαση των εκθέσεων ελέγχου των λογαριασμών όπου εξηγούνται επακριβώς τα διάφορα στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και ε, των ενεργειών της και να μπορέσει ε, να αποδείξει την ε, αποτελεσματικότητα του συστήματος και όχι μόνο σε από την οικονομική πλευρά. Η τελική έκθεση επικεντρώνεται στις παρατηρήσεις του Γενικού Διευθυντού και υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις οι οποίες κάπως μειώθηκαν το 2008 σε σχέση με το 2007 η εμβέλεια των επιφυλάξεων επίσης έχει μειωθεί από πλευράς αριθμού κρατών και προγραμμάτων. Ορισμένα θέματα που είχαν ε, ε, ανακύψει το 2008 έχουν ε, επιληθεί και υπήρξαν και ορισμένα λάθη. Σε 15 ε, τομείς ε, οι γενικές διευθύνσεις εξέφρασαν επιφυλάξεις και το συλλογικό όργανο ανέλαβε την ευθύνη αυτών των επιφυλάξεων που βασίζονται σε προγράμματα δράσης ε, ένας τομέας ε, ο οποίος ε, παρουσιάζει προβλήματα είχε εντοπιστεί ήδη στην έκθεση του 2007 από το ελεγκτικό συνέδριο και το 2008 η ευρωπαϊκή πολιτική προέβη σε ε, διάφορες βελτιώσεις ε, κατά 1,6 εκατομμυρίων ευρώ στους σχετικούς λογαριασμούς ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξε ότι ήθελε να μειώσει το ποσοστό των λαθών που ανήρχονται το 2007 σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ε, για το σύνολο των κρατών μερών και ε, η συνθετική έκθεση παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα διότι παρά τα πρώτα αποτελέσματα υπάρχουν ενδείξεις ότι η συλλογική στρατηγική δεν επαρκεί για να επιτευχθεί ο στόχος μειώσεως του ποσοστού ελέγχου, ε, του ποσοστού λάθους κάτω του 2%. Πρέπει να υπάρχει μία κοινή αποδοχή του ανεκτού ποσοστού λαθών, πράγμα το οποίο ίσως ισχύσει το 2010 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ε, για να προωθήσει τα θέματα. Και κυρίως για την έρευνα. Τώρα για την κοινή διαχείριση με τους φορείς του ΟΗΕ, αυτό είναι ένα θέμα ε, που εξετάζεται και του δίδεται ιδιαίτερη προσοχή. Η έκθεση του 2008 συμπεριλαμβάνει και διάφορα εγκάρσια θέματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Ένα από αυτά να αναφέρω μάλλον. Αυστηροί έλεγχοι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφεραν στο φω κάποιε ατασταλίε σε διάφορε πολιτικέ όσον αφορά τη διαχείριση πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι επιφυλάξει όσον αφορά τη διαχείριση κοινοτικών πόρων στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία οδήγησαν σε διευρυμένο συντονισμό μεταξύ των φορέων και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την υποστήριξη τη μεταρρυθμίσεω και των σχετικών προσπαθειών που καταβάλλονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα τα προβλήματα θα επιληθούν και ότι η διαχείριση όλων των πόλεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα λαμβάνει χώρα με αυστηρή συμμόρφωση στου κανόνε και διαδικασίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα δέχεται αδυναμίες μεγάλες συστημάτων και ατασταλίες από πλευράς αδίποτε εθνικής αρχής που χειρίζονται ευρωπαϊκούς πόρους σαν ένα μέρος της συνέχειας που θα δοθεί στην απαλλαγή, την έκθεση απαλλαγής του 2007 όσον αφορά την εφαρμογή των πόρων ε, είδατε μάλλον τα πορίσματα από αυτή την έκθεση που σας διαβάστηκαν. Κατακλείδη, εξότιμα μέλη. Αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να πετύχει θετική δήλωση εξοπιστίας. Αυτή η φιλοδοξία έχει θετικέ συνέπειε όσον αφορά το θεσμικό όργανο. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που ισχύει με τι διάφορε επιφυλάξει που συμπεριλαμβάνουν τι εκθέσει αιτησίων δραστηριοτήτων παρέχουν αναγκαίε διαβεβαιώσει ότι το 2008 οι πόροι που διατέθησαν για τι δραστηριότητέ μα χρησιμοποιήθηκαν για του σκοπού που αφιερώθηκαν και σύμφωνα με τι αρχέ τη ορθή οικονομική διαχείριση. Κύριε Πρόεδρε, εδώ κλείνω την παρουσίασή μου όσον αφορά την έκθεση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την έκθεσή τη για του εσωτερικού ελέγχου του 2008. Ο κύριο Γκρέι, ο ελεγκτή μα, είναι εδώ να παρουσιάσει σχετικά το θέμα αυτό και να σχολιάσει, αν το επιθυμείτε βεβαίω. Βεβαίως. είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Κάλλα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γκρέι. Για να διαλευκάνει τα όσα μα είπε μέχρι τώρα ο κύριο Κάλλα, να δώσω κάποιε εξηγήσει, Ο κύριο Γκρέι, ο οποίο λέει ο κύριο Γκρέι, ευχαριστώ και εσά και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού που μα δίνετε δυνατότητα να παρουσιάσετε τα βασικά στοιχεία τη ετησία εκθέσεω Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου που διενεργήθησαν το 2008. Όπως θα γνωρίζετε, διορίστηκαν επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου από 1η Ιουνίου του 2009 και έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στι προηγούμενε εκθέσει εσωτερικών ελέγχων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων μα του 2008 και δεν πληροφορίε τη συνέχεια που δίδεται στι συστάσει του εσωτερικού ελεγκτού. Εν γέννη, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εξέδωσε 93 εκθέσει ελέγχου, 36 από αυτέ αφορούν νέους ελέγχους και 51 εκθέσει αφορούν συστάσεις που απορρέουν από πρώτερου πρώτερους ελέγχους. Ο βαθμός αποδοχής από διάφορες υπηρεσίες των συστάσεων αυτών ήταν πολύ ε, υψηλό. 99,4% από τις 327 συστάσεις που δόθηκαν και καταρτίστηκαν από τις υπηρεσίες και σχέδια δράσεως σχετικά ο αντίκτυπο των συστάσεων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θελοποιηθούν τα σχέδια δράσεω και την ταχύτητα που θελοποιηθούν. Έχουμε και την Επιτροπή Προόδου Ελέγχων που ενημερώνουν του αρμόδιους επιτρόπους σχετικά με τις προόδου. Και αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό μέσο. Α εστιαστώ σε κάποια βασικά θέματα που αναφέρονται σε συμπεράσματα τη εκθέσεω. Σημαντικό θετικό συμπέρασμα πρώτα απ' όλα. Πρόοδος όσον αφορά τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Έξι συστάσεις βέβαια θεωρήθηκαν κρίσιμες σημασία το 2007. Αυτή τη φορά το 2008 είχαμε καμία. Και η έλλειψη ικανοποίηση, ή εν μέρη μη ικανοποιητικέ γνωμοδοτήσεις από έξι το 2007 ήταν 4 το 2008. Όμως πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όπω την χρηματοστηρική διαχείριση, όπου διαδικασίε για ανάκτηση, εντολέ ανάκτηση μπορούν να συντομευθούν και τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να βελτιωθούν. Διαδικασίε δημοπρασιών, προκηρύξεω διαγωνισμών μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα για να μην έχουμε συγκέντρωση στην αγορά. Δηλαδή να μην δίνουμε πολλέ συμβάσει σε λίγου που συμμετέχουν στου διαγωνισμού. Δεντρολογικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδαμε και ότι είναι πλήρε και στέρεο το σύστημα και θα πρέπει να ελέγχονται οι δράσεις που έχουν δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του 2010. Χρειάζεται προσοχή και πάλι στην έγκαιρη εφαρμογή κρισίμων και πολύ σημαντικών συστάσεων που απορρέουν από κάθε έλεγχο. Μια δραστηριότητα που καλείται όλου του τομεί και χαρακτήρισε το 2008 αφορούσε συστήματα τεχνολογίας IT, πληροφορική. Εκεί όλα εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα και τη σωστή λειτουργία του συστήματος του ψηφιακού. Ολοκληρωμένη προσέγγιση χρειάζεται και σωστή διαχείριση. Χρειάζεται βελτίωση και θα πρέπει να παρακολουθούμε και θέματα ασφαλείας όσον αφορά τα πληροφοριακά συστήματα, συστήματα που χρησιμοποιούν πληροφορική. Με χαρά άκουσα ότι η υπηρεσία ελέγχου λειτουργήσε καλά. Η αρμόδια επιτροπή στην έκθεση ποιοτικού ελέγχου δείχνει ότι οι έλεγχοι μα συμμορφώνονται με τι διεθνεί προδιαγραφέ. Επαγγελματισμό επεδείχθη στον εσωτερικό έλεγχο. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελέγχων καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία συμμορφωθήκαμε. Και επίση προβλέπεται και κατάρτιση για του ελεγκτέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε όλα τα πεδία. Για όλου του ελεγκτέ. Θέλουμε λοιπόν οι προδιαγραφέ αυτέ, τα πρότυπα, τα στάνταρ να παραμείνουν υψηλά. Στο μέλλον τι θα γίνει θα γίνονται έλεγχοι για χρηματοπιστωτικά και μη χρηματοπιστωτικά θέματα. Η εξολόγηση κινδύνου δείχνει ότι κίνδυνοι προκύπτουν και από μη οικονομικά θέματα. Νομικά, νομικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι που απορρέουν από κακή φήμη. Δεν πρέπει να μεληθούν και αυτοί οι κίνδυνοι. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο όσον αφορά την απαλλαγή του 2007 στον εισηγητή αντιπρόεδρο Jean-Pierre Audi. Ορίστε. Euh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα πρώτα μου λόγια είναι ευχαριστίες προς τις υπηρεσίες σας ε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαριστίες και προς εσάς για τις απαντήσεις που ετοιμάσατε και που μεταφέρατε ε, και διαβιβάσατε μάλλον στα μέλη της Επιτροπής μας δεχτήκατε σχεδόν όλες τις συστάσεις που κάναμε εμείς με κάποιες και σε αυτές θα επικεντρωθώ με κάποιες που αρνηθήκατε. Θα επανέλθω. Θέλω πάντως να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τη δουλειά σας. Και εκ μέρους μου κύριε Κάλλας, αν μη τι άλλο θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ που σας πρότεινε και πάλι για επίτροπο κυβέρνησή σας. Ήσασταν υπουργό στην Εστονία, πρωθυπουργό, ε, πρόεδρο τη Κεντρική Τράπεζα. Οπότε κύριε Κάλλας, ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που με έχει δοθεί ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας. Και βλέπω ότι έχετε προχωρήσει πάρα πολύ για όλα αυτά τα θέματα, τα οποία βέβαια δεν ξεσηκώνουν τα πάθη, αλλά είναι ζωτική σημασία για τη λειτουργία των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Κατόπιν τούτων, δεν θέλω να επανέλθω στα σημεία εκείνα με τα οποία είμαστε σύμφωνοι, οι υπηρεσίε της Επιτροπής και εμείς, αλλά θέλω να αναφερθώ στα σημεία εκείνα με τα οποία δεν συμφωνείτε. Πρώτα απ' όλα, η απαρίθμηση της ε, απαλλαγής. Στο σημείο 11 ζητήσαμε να ληφθούν υπόψη 33,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κράτη-μέλη σαν συντάξεις του προσωπικού. Εσείς σε αυτό δεν δίνεται απάντηση. Και όμως εμείς, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλουμε να δώσουμε την απαλλογή στους λογαριασμούς και ξέρω από τον συνάδελφο που είναι αρμόδιος για την απαλλογή ε, για το 2008 που ήταν, έχει φτάσει στο 36,9 και 4 μάλιστα. Οπότε γι' αυτό θέλω απάντηση σε αυτό το σημείο 11. Πάντα για το σημείο 11 έχουμε ζητήσει επίσης και μία μελέτη. Και τι μας λέτε εδώ, ότι δεν θα δώσετε συνέχεια στο έτοιμα μας αυτό, γιατί υπήρξε μία μελέτη παλιότερα η οποία είχε δείξει ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Μα η πρόταση δεν έλεγε είναι ή δεν είναι επικίνδυνο το χείρημα. Το θέμα είναι ότι οι συνταξιούχοι των κοινοτικών οργάνων και οι υπάλληλοι πρέπει να ξέρουν υπάρχουν τα χρήματα σε ένα συνταξιδιωτικό ταμείο. Αυτή τη διασφάλιση θέλουν. Θέλουν να το ξέρουν για να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ώστε οι επενδύσεις να γίνονται χωρίς ε, να τίθεται σε κίνδυνο το κεφάλαιο. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Στη σημερινή συγκύρια καταλαβαίνετε ότι η απάντησή σας δεν ε, ικανοποιεί. Στο σημείο 12 τώρα εμεί ρωτάμε γιατί το Γαλιλαίο και οι συμβάσεις του έγιναν, ε, που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου του 2007 δεν ελήφθησαν υπόψη. Ούτε εδώ πήραμε απάντηση. Στο σημείο 13 τώρα. Ε, απαντάτε ότι για τα κτίρια δεν θέλετε να τα λάβετε υπόψη. Εντάξει, μπορεί να είναι μικρότερη σημασία, αλλά παρόλα αυτά έχουμε κτίρια, τα οποία είναι καινούρια σχετικά. Και κάποια στιγμή θα χρειαστούν επιδιορθώσεις. Αν δεν έχουν προβλεφθεί αυτά τα χρήματα σαν επιδιορθώσεις, αν μη τι άλλο να μπουν στο αποθεματικό για τα κτίρια. Σημείο 14 για τους οργανισμούς, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε ότι έχουμε την πολιτική εξουσία πάνω στους οργανισμούς αυτούς. Απαντάτε μεν καταφατικά, αλλά πρέπει εδώ νομίζω να προσέξουμε περισσότερο η πολιτική εξουσία που έχουμε ε, σε αυτές τις κοινοτικέ υπηρεσίε να παγιωθεί. Στην παράγραφο 31 τώρα δεν θέλετε μελέτη για την ανεξαρτησία των εθνικών συστημάτων δίκησης για την ετήσια σύνοψη. Έχοντας πάει σε κάποιες από αυτές τις δικήσεις, όπου οι επικεφαλείς ορίζονται από τους ε, υψηλότερα στάμενους, τους ε, ιεραρχικά νότερους, η εξέταση της ανεξαρτησίας αυτών των δομών θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις αιτήσει αυτές ε, περιλήψεις στη διαδικασία απαλλαγή. Δηλαδή το Λεκτικό συνέδριο να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις αιτήσει ε, περιλήψεις ε, ξέροντας ότι μπορεί να βασιστεί σε ένα βαθμό γιατί είναι σύμφωνος με τις διεθνές προδιαγραφές. Οπότε λυπούμε που στην παράγραφο 34 εκεί που υπογραμμίζουμε την εφαρμογή του άρθρου 148.2 που λέει ότι είναι θεματοφύλακας βέβαια η Επιτροπή ε, λοιπόν, λέει λοιπόν εκεί ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τον Εθνικό Έλεγχο. Η συνεργασία αυτή γίνεται βέβαια με διάλογο, με σχέσεις ε, τεχνικές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επιχειρησιακά όμως θα έλεγα ότι η σχέση που έχουμε δεν χρησιμοποιείται αρκετά ενώ είναι κάτι που προβλέπεται από τις ηθίκες. Ανυπομονώ λοιπόν να ξέρω την άποψη του Λεκτικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την εφαρμογή της ηθίκης της Λισαβόνας πάνω σε αυτό το θέμα, μια που αυτή επιτρέπει στο Λεκτικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο να συλλέξει κάθε αναγκαία πληροφορία για να φέρει σε πέρος το έργο του, όσον αφορά τον έλεγχο δηλαδή των θεσμικών οργάνων. Συνεπώς εδώ έχουμε μία νομική βάση αρκετά ισχυρή, αρκετά πλούσια για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας τον έλεγχο και εφόσον δεν έχουμε τις εθνικές δηλώσεις που δεν υπογράφουν τελικά είτε πρωθυπουργοί είτε επικεφαλής, αν μη τι άλλο έχουμε κάποια τεκμηρίωση ποιότητας ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε τις διεθνείς προδιαγραφές ελέγχου. Τέλος, κάτι για την έρευνα. Σημείωσα την απάντηση που μας δίνετε που λέτε «Μα είναι η εφαρμογή των κανόνων, είναι κάτι περίπλοκο, αλλά έτσι είναι». Εγώ όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα για το θέμα της έρευνας να μπορούμε να έχουμε μία μελέτη, ένα έγγραφο τέλος πάντων, το οποίο να δείχνει ποια είναι η θέση του καθενός. Γιατί ε, αυτό που ακούμε εμείς, αυτό που φτάνει στα αυτιά μας είναι ότι ο τρόπο ελέγχου διαφέρει και καταλήγουμε στο πρόβλημα η εφαρμογή των κανόνων περίπλοκων. Έχουν σαν αποτέλεσμα να μας λένε οι διάφορες μονάδες ότι οι ελεγκτές που μπορεί να μην είσαστε εσείς, μπορεί να είναι αυτοί που πληρώνουμε απ' έξω, εξωτερικοί, δίνουν μια ερμηνεία στους κανόνες και τους υπολογισμούς για τις οικονομικές επιστροφές ε, τους κάνουν και οδηγούνται σε ποσά, το οποίο τελικά καταλήγουν σε ένα κλίμα απέναντι στα θεσμικά μας όργανα που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να διορθωθεί. Το θέμα δεν είναι να πλουταίνουν οι μεν και να φτωχαίνουν οι δε, είναι η εξοπιστία. Και αυτό είναι που φοβάμαι ότι πλήττεται εδώ. Θα ήθελα λοιπόν ένα τεχνικό αναγραφό από εσά, γι' αυτό το θέμα της έρευνας. Αυτά. Νομίζω ότι δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Χαίρομαι πάντως που εσείς ε, θέτετε σε εφαρμογή την επιθυμία του Πρόεδρου Μπαρόσο που ήταν να έχουμε μια θετική δήλωση αξιοπιστίας σε αντίθεση με το όσα το 2004, εσείς έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας και λέτε ότι είναι αυτός ο στόχος. Θετική ντάς. Πολύ σημαντικό αυτό, σε συνεργασία με το Ελεκτικό Συνέδριο, που στο κάτω-κάτω αυτή είναι η αποστολή του, όχι απλώς να δίνει μια δήλωση αξιοπιστία, αλλά να βοηθάει την Επιτροπή μας, να τη συνοδεύει, να τη διευκολύνει, προκειμένου να έχουμε θετική δήλωση αξιοπιστία. Χαιρόμαστε λοιπόν για αυτή τη δήλωση και ανυπομονούμε να δούμε τη συνέχεια των εργασιών σας για το 2007, μια που θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την απαλλαγή του 2008, όπου να είναι. Όσον αφορά την απαλλαγή του 2008, να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο, τον κύριο Κάλλας. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια σχετικά με το θέμα αυτό. Να προσθέσω κάποια στοιχεία στα ήδη υποθέτα από τον κύριο Ντί. Είχα τη χαρά να σας ακούσω, να ακούσω την παρουσίασή σας επανειλημμένα. Και σε αυτή την Επιτροπή και αλλού. Σας ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη παρουσίαση. Όσον αφορά το θέμα, το έτος 2008, όλα τα προβληθέντα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν από τους ομιλητές, πράγματι είναι ορθά. Θέλω να προσθέσω κάτι Πιστεύω ότι πράγματι η απόδοση, η αποτελεσματικότητα των λεκτικών συστημάτων βελτιώθηκε. Όμως υπάρχουν κάποιοι κρίσιμοι τομείς που παρουσιάζουν προβλήματα. Και εκεί θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις. Πρόβλημα 1. Επίπεδο σφαλμάτων. Σε επίπεδο 100 μελών. Το ποσοστό των σφαλμάτων σε επίπεδο 100 μελών. Κάτι το οποίο δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αναφέρομαι στην κατηγοριοποίηση των σφαλμάτων, την επαρκή κατηγοριοποίηση των σφαλμάτων. Σε ποιο βαθμό έγινε σφάλμα εκεί. Μέχρι το 2007, έχουμε το 2008, ένα σχέδιο 21 σημείο για την ανάκτηση πόρων και συναφείς δράσεις. Το ερώτημά μου, σε ποιο βαθμό πετύχατε όσον αφορά την ανάκτηση πόρων του 2006, όπου εκεί είχαμε 12% σφάλμα και το 2007, διότι συνολικά λείπουν 9 δις ευρώ. Σε ποιο βαθμό καταφέραμε να ανακτήσουμε τους πόρους όσον αφορά τα δύο έτη αυτά, αλλά και το 2008, δηλαδή 2006, 2007 και 2008. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι συζητήσαμε εκτενώς το πακέτο των 21 σημείων πέρσι στην ίδια αίθουσα. Οπότε διαρωτώ με πώς θα πήγε και κάτι άλλο. Οι εξωτερικές δράσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως αποκαλούνται. Όταν αναφερόμαστε σε αυτές, προφανώς γνωρίζουμε ότι είχαν προσημειωθεί κάποιοι πόροι για το συγκεκριμένο τομέα. Και καμιά φορά όταν υποβάλαμε ερωτήσεις λαμβάναμε απαντήσεις κάπως απροσδόκητες. Ίσως όχι μόνο από εσά κύριε Κάλλο, όχι από εσά και μόνο, αλλά μας είπαν ότι προφανώς δαπανήθηκαν τα χρήματα, αλλά ποτέ δεν ήμασταν σίγουροι σε ποιο βαθμό ήταν αποτελεσματική η χρήση των πόρων, κυρίως σε δράσεις που προσπαθούσαμε να εστιαστούμε στην καταπολέμηση της φτώχειας, παροχή βοήθειας, κυρίως σε περιοχές όπου υπήρχαν σειράξεις. Σε ποιο βαθμό υπάρχουν πόροι ακόμα εκεί. Σε ποιο βαθμό τα επενδυθέντα χρήματα μεταφράστηκαν σε καλύτερη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύτερη φήμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τα αναπτυξιακά, οι αναπτυξιακοί πόροι. Είχαμε προβλήματα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με τον ΟΗΕ. Σε κάποια φάση μας έλειπαν πληροφορίες όσον αφορά τις συνέπειες των επενδύσεων αυτών. Το κόστος κάθε χρόνο είναι δισεκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια ευρώ με συγχωρείτε. Θα θέλαμε να ακούμε περισσότερο για τα αποτελέσματα. Έρευνα. Συζητήσαμε εκτενώς την έρευνα. Εγώ έχω αναμειχθεί σε προγράμματα ερευνητικά υπό την επαγγελματική μου ιδιότητα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Με τον Κοπέρνικο. Όταν σκέφτομαι τον Κοπέρνικο έχω την εντύπωση ότι κανένας δεν τον δεν δίνει εντολή, να, δεν του δώσε εντολή του Κοπέρνικου, του πραγματικού Κοπέρνικου να ερευνήσει το πώς περιστρέφεται η γη γύρω από τον ήλιο. Δεν του είπε Κοπέρνικε ψάξτο και μετά τον πλήρωσε για τα αποτελέσματά του. Ξέρουμε όμως ότι άλλαξαν οι καιροί. Και τώρα έχουμε προγράμματα προχωρημένα, όπως το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Και ξέρουμε ότι τα χρήματα που δαπανίσαμε σε κάποιο βαθμό δεν ήταν όσο αποτελεσματικά θέλαμε, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Ποια είναι η άποψή σα για το θέμα αυτό. Τα συστήματα πληροφορικής, συστήματα IT. Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου για να δούμε κατά πόσο ήταν επιτυχής η προσπάθεια. Προφανώ είμαστε ικανοποιημένοι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε θετική αξιοπιστία αξιοπιστίας από πολλά κράτη-μέλη. Αλλά είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση μεταξύ των δηλώσεων αξιοπιστία. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι αυτές οι δηλώσεις δεν είναι εύκολα συγκρίσιμες. Ερώτηση. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό, μπορούμε να βελτιώσουμε τη συγκρισιμότητα των δηλώσεων αξιοπιστία των κρατών μελών, διότι καμιά φορά ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας λέει ότι κάποιες από τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές διότι τα κράτη-μέλη δεν παρέχουν τα σχετικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, όταν πηγαίνουμε στα κράτη-μέλη, εκεί μας λέγουν ότι υπάρχει πρόβλημα λόγω γραφειοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρεμφερεί επιχειρήματα. Ερώτηση. Θα ήταν δυνατόν. Εγώ είμαι σίγουρο θα ήταν δυνατόν. Θα ήταν δυνατόν να βελτιωθεί σε αυτό το επίπεδο συνεργασία. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσία σα. Για την παρουσίασή σα επίση. Και χαίρομαι που κρατήσατε τη θέση σας και παραμείνατε και στον ίδιο τομέα αρμοδιοτήτων και προσβλέπω σε μελλοντική συνεργασία μου μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ζήτησε το λόγο η κυρία Γκράσα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι καλό μήνυμα αυτό το οποίο μας μεταδώσατε και βέβαια αντιλαμβάνουμε ότι ακόμη έχουμε διάφορες δηλώσεις ε, αξιοπιστίες οι οποίες ε, δεν έχουν ε, κατατεθεί αλλά σε πολλά πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εργαστεί πολύ θετικά και αυτό εκφράζω εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε πάρα πολύ ενεργά και σας είμαστε ευγνώμονες. Ε, έχουμε ακόμη ε, ε, θέματα για τις χρήσεις 2004-2005 και υπάρχουν ε, και άλλες εκκρεμότητες και γι' αυτό θα ήθελα εδώ ε, να κάνω λίγες ερωτήσεις. Δηλαδή, τι προβλέψεις υπάρχουν για αποθέματα. Τι, ε, τι θεωρούμε σαν reportational risk υπάρχει για τις επικοινωνίες ένα απόθεμα για παραβιάσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν τομείς ε, στους οποίους τακτικά υπάρχουν προβλέψεις ενώ σε άλλους τομείς από το 2004 δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για, και κανένα απόθεμα για το ΕΚΟ, για το ε, ΕΤΚΟ και ε, υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν δαπάνες γιατί λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη μου ερώτηση, γιατί δεν έχουν γίνει καθόλου αποθέματα σε αυτούς τους τομείς. Μπορείτε να μου πείτε και να με βεβαιώσετε ότι δεν, χρειάζομαι, ε, δεν χρειαζόμαστε τέτοια αποθέματα και δεν πρόκειται να υπάρχουν λάθη ή δεν είναι κανείς αρμόδιος και δεν ευθύνεται για αυτά τα λάθη. Διότι νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε εμπιστευτούμε μόνο μερικό τα στοιχεία που μας δίνεται διότι δεν υπάρχουν κοινά μέτρα και σταθμά και ε, κανείς δεν καθορίζει ένα μέτρο το οποίο να ελέγχεται από τη Γενική Διεύθυνση και σύμφωνα με το οποίο να γίνονται και οι έλεγχοι. Ε, άκουσα για τους ελέγχους της ΕΤΚΟ ότι ε, αφιερώνεται πολλές σελίδες στην ΕΤΚΟ Πρόκειται για πολύ σημαντικές συστάσεις τις οποίες έχετε διατυπώσει και θα ήταν καλό να ξέρουμε παραδείγματο χάρη ε, ποιες είναι αυτές ε, οι συστάσεις και εσείς ε, πώς αξιολογείτε τις δαπάνες της ΕΤΚΟ και τις δαπάνες οι οποίες αποδίδονται στον ΟΗΕ. Στη συνθετική έκθεση λέγεται ότι έχουν δαπανηθεί 3 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά από ποιο ποσό, τι θα έπρεπε να έχουμε προβλέψει ε, ποιος είναι ποιο είναι το ποσό βάσεω το οποίο θα έπρεπε να έχουμε ε, περιλάβει στα αποθέματα διότι και η όλα ξέρω ότι ε, έχει ορισμένες προβλέψεις αλλά υπάρχουν υπάρχουν πολλοί τομείς όπου οι μετρήσεις δεν είναι σαφείς. Ή στην ε, ε, Ρουμανία υπάρχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα αλλά οι πληρωμές έγιναν το, από το 2007 το 2008 για τις προενταξιακές δαπάνες ε, σε τι οφείλεται αυτό σε αυστηρούς ελέγχους τι έγινε πριν από το 2007-2008 στις χώρες αυτές δεν υπήρχαν έλεγχοι γιατί λέγεται ότι υπήρχε πρόβλημα με το δικό σύστημα το 2007 στην ε, Βουλγαρία τα ποσά αποδεσμεύτηκαν το 2008 έγινε θαύμα ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ό,τι δεν ε, χρειάζεται ε, μπορεί ε, να εφαρμοστεί ε, πιο γρήγορα στα κράτη-μέλη από ό,τι σε αυτήν. Δηλαδή αυτή μπορεί να καθυστερεί και τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμορφώνονται άμεσα. Ε, έχουμε αποθέματα και για προενταξιακή βοήθεια και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ανδρέας είναι επόμενος αγορητής. Κυρία Ανδρέασεν μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάλλας και κύριε Γκρέι για την παρουσίασή σας, τις εκθέσεις σας στην ετήσια ε, έκθεση ε, δραστηριοτήτων λέγεται ότι έγινε ποιοτική αξιολόγηση και ότι συνάδει με τις ε, απαιτήσει των εσωτερικών ελεγχών θα ήθελα να ξέρω ποιος έκανε αυτή την αξιολόγηση ποιότητος, ποιος την πλήρωσε και αν η εταιρεία ή η οργάνωση που έκανε αυτή την αξιολόγηση δέχεται ε, ο τωρινός εσωτερικός ελεγκτής να είναι ο πρώην δηλαδή ο ίδιος να ελέγχει τα συστήματα τα οποία κατήρτισε πριν από δύο-τρία χρόνια. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να διευκρινίσω είναι ότι στις αιτήσιες δηλώσεις ε, στην έκθεσή σας λέγεται ότι έχετε ε, ε, λιγότερες επιφυλάξεις. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των λαθών έχει μειωθεί ή το ποσοστό των ελέγχων έχει μειωθεί και επίσης θα ήθελα να ξέρω πόσο καθορίζεται ε, τα τις δημοσιονομικές διορθώσεις τις οποίες πρέπει να κάνετε για παρελθούσες χρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Χαζημαρκά, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ εν ονόματι της πολιτικής μου ομάδος να ευχαριστήσω τον Επίτροπο γιατί δεν ήταν πάντοτε εύκολη η κατάσταση και γι' αυτό πρέπει εγώ να σας πω ότι η εργασία την οποία κάνετε είναι εξαιρετική και θέλω να σας συγχαρώ για αυτό. Πράγμα το οποίο αποδειχνεί ότι στην λεπτομέρεια και στην επιμονή οφείλεται και η αμοιβή. Διότι έλαβα τα National Summaries με την αγγλική έκφραση και ξέρετε ότι πάντοτε ζητούσαμε τις Management Declarations σε αυτές τις περιλήψεις. Δεν έχουμε επιτύχει το στόχο μας αλλά έχουμε προχωρήσει και εδώ πολύ χάρη στη δουλειά σας. Γι' αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω, πράγμα όμως το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας και ότι τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να ενθαρρυνθούν, δεν θα πω να υποχρεωθούν, να μας δίνουν καλύτερες και πιο ακριβείς πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Κάλλας, διότι του ετέθησαν διάφορες ερωτήσεις και ακούστηκαν διάφορα σχόλια απευθυνόμενα προς αυτόν. Έχετε το λόγο κύριε σε Ευχαριστώ αξιότιμα μέλη για τις ερωτήσεις σας και θα ήθελα να σας πω ότι ευθύς εξ αρχής στην αρχή μάλλον θα έχουμε πολύ πιεστικό πρόγραμμα διότι ο πρόεδρος Κλάους υπέβαλε τις συνθήκες της Αβώνας. Οπότε θα μας πιέσει ο χρόνος. Θα βασιστούμε λοιπόν σε αυτό το γεγονός, σε αυτές τις νέες εξελίξεις. Uh, uh, Αρκετοί λοιπόν θα έχουν αρκετέ δυνατότητες να εμφανιστούν στην Επιτροπή σας. Και σύντομα μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις ερωτήσεις που μου απευθύνθησαν, όσον αφορά τα θέματα λογιστικής που έθεσε ο κύριος Σοντή, πιθανότατα πιο αρμόδιος ο Φίλιπ Ταβέρν είναι να απαντήσει που είναι ο επικεφαλής του λογιστικού τμήματος και μπορεί να δώσει λεπτομερέστερες απαντήσεις. Γενική απάντηση όμως. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν σε εκθέσεις. Υπάρχουν αριθμοί, στοιχεία για το Γαλιλαίος, για τα κτίρια, για τις εγγυήσεις, Το θέμα είναι πώς αντικατοπτρίζονται αυτά τα στοιχεία, αυτοί οι αριθμοί στα λογιστικά. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες για λογιστική που διέπουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό, υπάρχουν τα στοιχεία. Μπορούν να εξεταστούν. Η απάντηση είναι ότι οι διεθνείς λογιστικοί κανόνες προβλέπουν κάποια πράγματα και εμείς συμμορφωνόμαστε για τις υπηρεσίες και τον έλεγχο αυτών. Το συζητήσαμε επανειλημμένα στην Επιτροπή. Και υπάρχει πράγματι πρόβλημα. Οι υπηρεσίες φυτρώνουν παντού, οι ρυθμιστικέ υπηρεσίες φυτρώνουν παντού σαν μανιτάρια. Και είναι ανεξάρτητοι φορεί νομικά πρόσωπα. Και πρέπει να παίρνουν απαλλαγή όπως παίρνει απαλλαγή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι στο ίδιο επίπεδο, Όπω και εμεί. και ελέγχονται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για να αποφύγουμε προβλήματα. Αυτό είναι ένα θέμα. Κάθε υπηρεσία έχει τη δική της νομική βάση και είναι υπόλογη άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από κράτη-μέλη και τα αποτελέσματα του ελέγχου παρέχονται σε αυτούς. Δεν υπάρχει ε, πληροφόρηση που πηγαίνει προς τα εμάς και κεντρική οικονομική διαχείριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή όσον αφορά τους τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών. Έρευνα Πολλοί αναφέρθηκαν στην έρευνα. Ποια είναι η ιστορική ροή των πραγμάτων. Όταν ξεκινήσαμε, η έρευνα ήταν η πλέον ευάλωτη περιοχή στον αυτά τα σφάλματα. Επεκρίθη τα μάλα στην Επιτροπή Ενέχου Προπολογισμού, στην πρώτη απαλλαγή μας. Ο τομέας της έρευνας είχε τα περισσότερα σφάλματα. καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες ελεγκτικές και ενισχύσεως των ελέγχων. Και απαιτούμε επιστροφή χρημάτων. Και δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τι έρευνε, Δηλαδή, γραφειοκρατία, ποιοι κανόνες ισχύουν και ούτω καθεξής. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Θέλουμε να ακούσουμε προτάσεις για πλούστευση των κανόνων όσον αφορά την έρευνα. Ταυτόχρονα, Υπάρχουν κάποιες απαιτήσει. Και θα πρέπει να αποδεικνύεται το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Πραγματικά πώς χρησιμοποιούνται, αν χρησιμοποιούνται σωστά, ορθά, σύμφωνα με τους κανόνες. Πάντα υπάρχει αυτό το δίλημα. Ο κύριος Λιμπεράτσκι το έθεσε σωστά. Κανείς δεν προέβλεπε τα αποτελέσματα της πραγματικής έρευνας. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όπως και σε άλλα προγράμματα σε, άλλου τομεί άλλους μπορείς να προβλέψεις κάποιο αποτέλεσμα. Στην έρευνα δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να πεις τώρα θα πετύχεις μια θερμοπυρηνική αντίδραση, ο αντιδραστήρας θα είναι έτοιμος για τη συγκεκριμένη θερμοπυρηνική αντίδραση σε τόσα χρόνια. Είναι αδύνατον αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη βάση για την αξιολόγηση της χρήσης των πόρων για την έρευνα. Υπάρχουν κάποια έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι χρησιμοποιούνται σωστά οι πόροι και δεν εξαφανίζονται. Πώς πετυχαίνουμε τη σωστή ισορροπία. Hm. Το συζήτησα με τον Γιάννου Πότερσνικ, το συνάδελφο το θέμα, επανειλημμένα. Και αυτός ανησυχεί, ανησυχεί και απογοητεύεται και η επιστημονική κοινότητα γιατί είναι άκαμπτη η προσέγγιση μας ο ανεκτός κίνδυνος. Το επίπεδο των σφαλμάτων θα πρέπει να αποφασιστεί. Αλλά είναι περίπλοκο πολιτικό θέμα. Εξωτερική βοήθεια. Το ίδιο. Ενισχύσαμε. Πώς να το πω, τις απαιτήσει μας όσον αφορά την χρήση των πόρων για την εξωτερική βοήθεια. Πολύ περίπλοκος τομέας, το ξέρετε. Επί σειρά ετών έχετε διεξάγει ακροάσεις. Έχουν παρουσιαστεί επίτροποι που αναφέρθηκαν στο θέμα, αλλά είναι πολύ ευαίσθητος τομέας, πολύ πολιτικός τομέας. Χρηματοδοτούμε πάρα πολλά προγράμματα διεθνών οργανισμών, κυρίως μέσω του ΟΗΕ. και άλλων οργανισμών που εξαρτώνται από τον ΟΗΕ. Και πρέπει να αξιολογούμε πώς χειρίζονται τα χρήματα. Έχουμε κριτήρια γι' αυτό. Πώς συμμορφώνεται η χρήση των χρημάτων με τις απαιτήσει μας. Αλλά για συγκεκριμένα προγράμματα είναι επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση. Ακολουθούμε μια γενική προσέγγιση. Μπορούμε να μπούμε σε κάθε πρόγραμμα δύσκολο να συμφωνήσουμε με αυτούς τους φορείς. Οι ίδιοι οργανισμοί. Εγώ πήγα στον ΟΗΕ, ζήτησα περισσότερα, περισσότερες πληροφορίες, καλύτερη συνεργασία, μας το υποσχέθηκαν. Το εξετάσαμε στην έκθεση προόδου ελέγχου. Το συζητήσαμε και με αντιπροσωπείε του ΟΗΕ. Υπάρχει προθυμία συνεργασίας. Υπάρχει προθυμία για ανταλλαγή πληροφοριών. Χρειάζεται όμως περισσότερη συνεργασία. Χρειάζεται σωστή προσέγγιση. Χρειάζεται σωστή ισορροπία. Ο ΙΕ. Τώρα, κίνδυνοι για τη φήμη, για την εικόνα μας προς τα έξω. Α, πρώτα σφάλματα. Ποια σφάλματα διορθώθηκαν. Το περίφημο 12% που ανέφερε ο αξιότιμος συγγητής βασιζόταν σε κάποια επέκταση δειγματοληπτική των γραφημάτων. Τα δείγματα αποτελούσαν βάση. Εγώ δεν αμφισβητώ τη μεθοδολογία. Πώς να δουλέψει κανείς χωρίς προβολή στατιστική. Διορθώθηκαν όμως τα δείγματα. Ξεμπερδέψαμε το 12% σχεδόν του. Αυξήθηκε η ανάκτηση Στη συνοπτική έκθεση φαίνονται τα στοιχεία. Περίπου 3 δισεκατομμύρια το 2008. Ανάκτηση. Η κυρία Γκρέσλε ρώτησε ποιο ποσοστό απολειών ανακτήθηκε. Χρησιμοποίησα εγώ κάποιο στοιχείο τελικό αποτέλεσμα κατανοητό της πάση. Τουλάχιστον όσων έχουν κάποια γνώση λογιστικών. Είναι οι απώλειες στα λογιστικά. Τα στοιχεία στο παράρτημα 6. Βλέπετε. Σύνοψη. Το 2008 έχασαν 18.380.363 ευρώ και 22 cents. Αυτά χάθηκαν. Πάνε. Πριν από κάνα δύο χρόνια ήταν 60 εκατομμύρια, αλλά τώρα είναι μικρό το ποσό. Του χρόνου μπορεί να ξαναπάει στα 60 εκατομμύρια. Λογιστικά είμαστε πάρα πολύ ακριβείς. Τελειώσαμε. Πάει. Φύγανε τα 18 εκατομμύρια. Ξεχάστε τα. Και όπως βλέπετε, αυτό το ποσό πραγματικών απολειών είναι αρκετά μικρό. Ερώτηση εκτός μικρόφωνου, διερμηνής δεν την ακούμε. Απάντηση. Κάθε χρόνο διαγράφουμε κάτι από τον ισολογισμό μας. Μπορείτε να τα δείτε αυτά. Αν έχετε συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να την καταγγείλετε. Μπορεί να την καταγγείλει, να προσπαθήσει να ανακτήσει τα χρήματα, τα κάνει όλα αυτά, γίνονται διορθώσει εγγράφων, στοιχείων, χρήματα επιστρέφουν. Κάνει του υπολογισμού σου και τελικά χάνει οριστικά κάποιο ποσό που δεν ανακτάται ποτέ. Αυτό ανέφερα πριν. Τώρα, ετήσιε εκθέσει δραστηριοτήτων και σχετική συνοχή είναι προφορικά έγγραφα, λέει ο μιλητή και δεν είναι πολύ ακριβή από πλευράς αριθμητικών στοιχείων. Αυτά τα χρόνια κάναμε προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούμε να το αποδείξουμε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε πολλά για να ομαδοποιήσουμε τα κείμενα και τα στοιχεία και τις κατευθυντήριες γραμμές που γίνουμε στους γενικούς διευθυντές. Πώς να βάζουν κάποιο ποσά και αποθεματικό κλπ. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη σύγκριση των εγγράφων έτσι. Καλύτερη σύγκριση των παρουσιάσεων. Βελτιώνονται τα πράγματα. Όσον αφορά οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους για τη φήμη μας, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη έχουν πολλά, πολλούς κινδύνους να αντιμετωπίσουν αφορά τη φήμη τους και την εικόνα τους. Πώς γίνεται η σύγκριση αυτών των κινδύνων όμως. Συζητήθηκε αυτό στην Επιτροπή Πρόοδου Ελέγχου επανειλημμένα. Καταλήξαμε σε κάποιο προσανατολισμό. Αυτή η κίνδυνοι για τη φήμη που προκύπτουν από τις ειδικές εκθέσεις, οι έρευνες, πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και στις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου. Αλλά τώρα να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το γενικό τοπίο των κινδύνων για την εικόνα μας, για τη φήμη μας, είναι σχεδόν ανέφικτο. Τεράστιο έργο. Δύσκολο θέμα. Συμφωνώ μαζί σας. Μπορούν κάποιοι κίνδυνοι να είναι πολύ υψηλότεροι για, από, όσον αφορά τη φήμαζα είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι κάποιοι οικονομικοί κίνδυνοι. Όσον αφορά την αξιολόγηση την ποιοτική, η APMG έκανε την αξιολόγηση. Ποιο έκανε την ποιοτική αξιολόγηση? Ernst Young, ναι. <laughs> Συγγνώμη. Πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τα χαράς να παρουσιάσουμε τα απορίσματα. Παρουσιάστηκε στο κοινό όταν και όταν γράφω. Είδαμε ισχυρά σημεία και αδυναμίες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Υπήρχαν και κάποιε επικρίσεις, τα περισσότερα θετικά βέβαια, όλα είναι ανοιχτά, διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλους. Σύγκρουση συμφερόντων. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι ο υπεύθυνο εσωτερικό έλεγχο πριν ήταν επικεφαλή του λογιστικού τμήματο. Δεν νομίζω υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η κυρία Αντρεάσεν έθεσε ένα ερώτημα. Όσον αφορά την επιφυλακτικότητά μας, προσπαθήσαμε να δώσουμε προσανατολισμό στους γενικούς διευθυντές όσον αφορά την προσέγγιση πρέπει να ακολουθούν. Και αν θυμόσαστε, στην αρχή της θητείας αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθήσαμε να δώσουμε πληροφορίες. Εμείς θέλαμε να είναι τίμιες οι πληροφορίες, να αντικατοπτήσουν πληροφορίες την πραγματικότητα. θα θυμούνται τα μέλη ότι η πρώτη επίκριση ήταν ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα κράτη-μέλη, για τις επιφυλάξεις. Δεν κατονομάζονται κράτη-μέλη. Βλέπετε ότι αντικατοπτήσει την κατάσταση των διαφόρων κρατών μελών. Οι εκθέσει ετησίων δραστηριοτήτων αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα όλο και περισσότερο. εθνικές δηλώσεις και αιτήσιες συνοπτικές εκθέσεις. Συζητήθηκε εκτενέστατα στην Επιτροπή Ενέχου Προπολογισμού το θέμα επί σειρά ετών. Και θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, πιστεύω. Εγώ ήμουν παρόν στην αρχή της θητείας μου αυτής που λύγει τώρα ήμουν απεπισμένος όσον αυτό το θέμα των εθνικών δηλώσεων. Ήμουν ενθουσιώδης και εξακολουθώ να τις θέλω. Ίσως όμως τώρα να είναι πιο ισορροπημένη η θέση μου. Οι εθνικές δηλώσεις δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Δική μας δουλειά είναι. Σε κεντρικό επίπεδο να γίνεται η διαχείριση. Οι αιτήσεις συνοπτικές εκθέσεις ετοιμάζονται. Δύο χρόνια γίνεται αυτή η δουλειά και υποβάλλονται τα κάτι μελη Βελτιώνεται συνεχώς η κατάσταση. Συνεργάζομαι με τις χώρες που εθελοντικά υπέβαλαν εθνικές δηλώσεις. Και χαίρομαι που συνεργάζομαι μαζί τους, κυρίως με τις κάτω χώρες που ξεκίνησαν. Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, που έδωσαν εθνικές δηλώσεις. Διαφέρουν μεταξύ τους όμως. Πολύ και προσπαθούμε να δούμε πώς οι εθνικές δηλώσεις μπορούν να βελτιωθούν. Θα πρέπει λοιπόν για να βελτιώσουμε την κατάσταση να ρυθμίσουμε πολλές λεπτομέρειες και να διευρύνουμε το πεδίο των εθνικών δηλώσεων, να χρησιμοποιούνται περισσότερο εθνικές δηλώσεις. Ο στόχος είναι αυτός που ανέφερε ο κύριος Σοντή. Η δήλωση αξιοπιστίας είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται δυσκολότατα. Πρέπει όμως να έχουμε και ιδεώδη, να είμαστε ιδεαλιστές, να θεωρήσουμε ότι μπορεί να βελτιωθούν τα πράγματα και να απαλλαγούμε από την αρνητική εικόνα που έχει δήλωση αξιοπιστίας. θα πρέπει τελικά να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια τόσο ώστε να λυθεί το θέμα των δηλώσεων εξοπιστίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, κύριε Επίτροπε Κάλλας. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, ας πάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την παρουσίαση της μελέτης του 5 Ιουνίου για τη διαχείριση, την κοινή διαχείριση. Οι αιτήσει συνόψει στο πλαίσιο τη μεμερισμένη διαχείριση αξιολόγηση, μελλοντική πορεία και ενδεχόμενη θυσιμότητα έλεγχο. Έστερ πρώτος που θα πάρει το λόγο. Η κυρία που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη για την ε, μελέτη αυτή. Θα ήθελα λιγάκι να θυμηθούμε ποιο ήταν το πλαίσιο για τις ετήσιες συνόψεις να καταλάβουν και καινούργοι εδώ. Πρόκειται λοιπόν για συνόψεις όσον αφορά την κοινή διαχείριση είναι δηλώσεις, αυτές οι δηλώσεις είναι μια πιο πρόσφατη εξέλιξη, το είχαν ζητήσει πολύ για την περίοδο 2007-2013. Προχωρήσαμε περισσότερο, ζητήσαμε πέρα από τις συνόψεις για την επιμερισμένη διαχείριση και μια πολιτική ευθύνη, μια διάσταση πολιτικής ευθύνης να συμπεριληφθεί εκεί. Και ο Επίτροπος είπε ότι σε θελοντική βάση ναι, μπορεί κάλλιστα να γίνει. Εξάλλου είναι κάτι που και σε εθνικό επίπεδο στη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλάβαμε ότι το θέλανε ήδη από το 2003. Τελικά συμφωνήθηκε να υπάρχει αυτή η ετήσια σύνοψη και πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό τη στιγμή που το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αυτή ζητάει επίμονα να έχει τις εθνικές συνόψεις. Θα δούμε πώς θα γίνει στην πράξη με αυτές τις ετήσιες συνόψεις. Εξού και η μελέτη Ανέλαβα να δω λοιπόν στη μελέτη μου αυτή πώς θα λειτουργήσει το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως όλους όσοι συνεργάστηκαν για τη μελέτη αυτή που πιστεύω ότι, είναι μια... ότι έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την απαλλαγή και όσον αφορά τον επόμενο προπολογισμό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διαβάσει την μελέτη αυτή. Από εκεί και πέρα οι ίδιοι οι ερευνητές μπορούν να μας πούνε περισσότερα για την μελέτη. Ωραία. Δίνω τότε το λόγο ευθύ αμέσω στον ε, αρμόδιο για αυτό το θέμα. Παρακαλώ που συνεργάστηκε δηλαδή τον ερευνητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Ειλικρινά έχουμε κάποια πρακτικά προβλήματα εδώ, τεχνικά προβλήματα με την παρουσίασή μας, οπότε χωρίς εικόνα θα σας πούμε τα της μελέτης. Παρακολουθήστε από το γραπτό να παρακολουθήσετε την παρουσίασή μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Όντως ήμουν επικεφαλής της μελέτης με τον συνάδελφό μου, Μίρισκραφ, θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Είναι μελέτη που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου και συμπληρώθηκε πριν από έξι μήνες περίπου, ολοκληρώθηκε. Πριν μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης μας και τα συμπεράσματα, θα ξεκινήσω με το πλαίσιο όσον αφορά την αρχιτεκτονική λογιστική της Επιτροπής και των κρατών μελών. Το άρθρο 274 της συνθήκης λέει ότι είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του προπολογισμού. Συγχρόνως όμως τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το σκοπό. Ας δούμε το πρώτο τμήμα του άρθρου πρώτα και ας το δούμε στο θεσμικό πλαίσιο. Αν κοιτάξετε τη διαφάνεια αριθμός 3, κάτω βλέπετε τους γενικούς διευθυντής που ετοιμάζουν έκθεση δραστηριοτήτων και η δήλωση αξιοπιστίας δίνεται από τον Γενικό Διευθυντή. Και σε επίπεδο επιτροπής οι δραστηριότητες παίρνουν μαζί στα συμπεράσματα. Όπως γνωρίζετε, το έγγραφο αυτό πηγαίνει στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών σαν στοιχείο για την απαλλαγή. Αυτό είναι στη μεσαία γραμμή. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα κατάλληλο επίπεδο φερεγγιότητας, πρέπει να έχουμε επιδόσεις σε κάθε επίπεδο οι ελεγκτικές προσπάθειες που γίνονται και σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου και σε επίπεδο υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά σε επίπεδο ελεγκτικού συνεδρίου. Και πάλι κοιτώντας στις διαφάνειες. Το σύστημα δεν δείχνει τόσο κακό, όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επίσης 80% περίπου του προπολογισμού είναι στα χέρια των κρατών μελών. Αυτή η εικόνα έχει να κάνει με το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο. Οπότε πρέπει να δούμε κάπως γρήγορα και τα εθνικά επίπεδα. Και το εθνικό επίπεδο περιγράφεται στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν κυρίως τρεις παράγοντες όσον αφορά την αλυσίδα σε εθνικό επίπεδο του ελέγχου υπάρχει η πιστοποίηση και μερικές φορές έχουμε και διάμεσα σώματα. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχει και από κοινού ευθύνη και σύνθετες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργάνων. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της κανονικότητας των λογαριασμών. Ε, τα διάφορα όργανα ετοιμάζουν ε, έγγραφα τα οποία οδηγούν τελικά στην δήλωση αξιοπιστίας σε διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχει εσωτερικός έλεγχος. Υπάρχουν επίσης τα διαχειριστικά προγράμματα από το άλλο επίπεδο. Όλα μαζί βασίζονται στα... Όλα αυτά μαζί μάλλον οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου και τις αιτήσιες συνοψίσεις. Βλέπετε εδώ τον τίτλο Annual Summaries. Όμως οι συνόψεις αυτές δεν έχουν πολιτικές επιπτώσεις. Περιορίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά και καθαρά πληροφορίες όσον αφορά τη διαχείριση. Αυτός λοιπόν είναι και ο κρίκος που λείπει ανάμεσα στους λογιστικούς ελέγχους σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, η μελέτη μας είχε να κάνει με τις αιτήσει συνόψεις. Α δούμε ποιο είναι ο νομικός ορισμός. Θα τον δείτε στην επόμενη διαφάνεια. Οι αιτήσει συνόψεις ρυθμίζονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό. Στο άρθρο 53β λέει ότι οι αιτήσει συνόψεις θα παράγονται στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο και μετά έχουμε και άλλες πιο συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά τις εφαρμοστικές διατάξεις. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνονται οι συνόψεις αυτές από το κατάλληλο όργανο που ορίζεται. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι έχουμε δύο τμήματα στις αιτήσεις συνόψεις. Ένα που έχει να κάνει με τους ελέγχου και ένα που έχει να κάνει με τις δηλώσεις. Συνεπώς, άπαξ και γνωρίζουμε ποιο είναι το θέμα της μελέτης μας ή της συνόψης, λοιπόν, μπορούμε να πάμε και στον στόχο μας. Γυρίστε σελίδα και δείτε την επόμενη διαφάνεια. Η στόχοι μας ήταν εξής. Από ό,τι φαίνεται η οθόνη δουλεύει, λέει ο μιλητής. Σε λίγο θα μπορούμε να σας δείξουμε και εικόνα των όσων λέμε. Okay, now it's, it's more readable. Um, όπως είπα λοιπόν, η στόχη μας ήταν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουμε την συμμόρφωση και τις επιπτώσεις των ε, ετησίων συνόψεων. Ιδιαίτερα συγκρίνοντας με τις δηλώσεις εθνικής διαχείρισης. Δεύτερος στόχος ήταν να κάνουμε συστάσεις για βελτίωση. πώς πετύχαμε τους στόχους μας και ποια ήταν η προσέγγισή μας. Αυτά τα βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια τώρα. Έχουμε την ανάλυση των συνόψεων για το έτος 2007 και μετά ε, κοιτάμε την ε, επεξεργασία για τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναλύουμε τι υπάρχουσες αξιολογήσεις πρώτα απ' όλα για να αποφύγουμε επικάλυψη. Και μετά μιλήσαμε με διάφορους ανθρώπους κλειδί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στείλαμε μάλιστα και ερωτηματολόγια σε όλα τα κράτη-μέλη για να δούμε ποιο είναι ο αρμόδιος, ποιο όργανο είναι αρμόδιο για την παραγωγή των ε, ετησίων συνόψεων. Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία με διάφορους και με υπηρεσίες από όλα τα κοινωτικά όργανα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν σε τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους οργανισμούς ελέγχου. Και τέλος είχα, θέλαμε και μια τελική επιβεβαίωση, οπότε ζητήσαμε από πυρογνώμονες να βοηθήσουν, να ξανακοιτάξουν δηλαδή το σχέδιό μας, το σχέδιο της μελέτης μας και να μας πούν τη γνώμη τους για τη μελέτη μας. Η μελέτη μας λοιπόν καλύπτει τέσσερις τομείς, κύρια. Τις διδικασίες, τις επιπτώσεις και τη χρησιμότητα των ετησίων συνόψεων όσον αφορά τη δήλωση εξοπιστίας. Θέλω να σας παρουσιάσω λοιπόν τα συμπεράσματά μας και τις συστάσεις μας για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Πρώτον, διαπιστώσαμε ότι η νομική βάση για τις ετήσιες συνόψεις είναι μάλλον ισχνή. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να κάνει το κείμενο όσο γίνεται καλύτερο βάζοντας μια διάκριση ανάμεσα στα υποχρεωτικά στοιχεία και στα, σε εθελοντική βάση, προαιρετικά στοιχεία. Επίσης συμπεράναμε ότι η Επιτροπή έχει κοιτάξει και τα τεχνικά ζητήματα. Όμως, σκεφτήκαμε ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής ήταν πολύ περιορισμένες. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές, το σημείο με αυτό, το σχετικό, εμείς διαπιστώσαμε ότι ήταν ξεκάθαρες, απλές και κατανοητές. Συγχρόνως όμως υπήρξαν και άλλες εκδοχές οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των ετησίων συνόψεων. Έπειτα υπήρχαν και τα μη υποχρεωτικά τμήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το θέμα των οργάνων που είχαν ε, εντολή ελέγχου. Το επόμενο έχει να κάνει με τις αντιδράσεις των κρατών μελών όσον αφορά το προαιρετικό σκέλος. Εμείς διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη αντιδράσεων από τα κράτη-μέλη που θα τα δείτε εδώ στη διαφάνεια. Συνεπώς βγάλαμε το συμπέρασμα ότι λίγες μόνο χώρες μέλη ακολούθησαν την ε, διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύνολο των τμήματων. Κάποια κράτη δήλωσαν απλώς ότι δεν υπάρχει συστηματικά κάποια διαπίστωση ή ότι δεν υπάρχουν αντιφάσεις στα στοιχεία που δίνονται. Κάποιες χώρες, από την άλλη, περιορίζουν την ανάλυση τους σε έναν κατάλογο μόνο ευρημάτων. Και τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν βρήκαμε τίποτα που να θεωρούμε ότι ικανοποιεί τους στόχους. Ο κύριος λόγος που δεν θέλουν να βάλουν προαιρετικά στοιχεία είναι η άρνηση των ε, οργάνων που έχουν οριστεί για αυτή τη δουλειά. Επόμενη διαφάνεια έχει να κάνει με τη νομική εκπροσώπηση των επιλεγμένων οργάνων. Πρώτα απ' όλα ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστεί μία νομική βάση. Επίσης διαπιστώσαμε ότι η εκπροσώπηση ήταν μάλλον σε χαμηλό επίπεδο. Μερικές φορές ήταν δύσκολο ακόμα και να εντοπίσουμε ποιος υπογράφει την ετήσια σύνοψη. Δεν ξέραμε ποιος την έχει υπογράψει. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ορισμένα όργανα ήταν μια αρχή Πρόκειται δηλαδή για ένα μπέρδαμα εδώ πέρα ελέγχου και διαχείρισης. βασισμένο λοιπόν στα βρέματα αυτά, καταλήξαμε σε κάποιες συστάσεις. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι η εφαρμογή των συστάσεων αυτών δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Οι συστάσεις λοιπόν είναι εξής. Πρώτον, όσον αφορά την νομική βάση στο δημοσιονομικό κανονισμό, πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν ε, σε κατάλληλο πολιτικό επίπεδο εκπροσώπηση τα κράτη-μέλη. Συστήνουμε επίσης, επίσης ότι πρέπει να αποτελούν οι αιτήσει συνόψεις μέρος της αιτήσιας δήλωσης αξιοπιστίας και να πρόκειται για σώματα που έχουν ευθύνες, έχουν συγκεκριμένη νομική ευθύνη. Πρέπει να υπάρχει επίσης ρητή μνήα για το ποιο υπογράφει. Να μπορούμε να εντοπίσουμε δηλαδή τελικά Ποιο είναι ο υπεύθυνο για την ετήσια σύνοψη. Έναν άλλο τομέα που καλύπτει η μελέτη μας ήταν οι επιπτώσεις και η προστιθέμενη αξία των ετήσιων συνόψεων. Ευρήματα. Το κύριο είναι ότι πρόσθετη αξία των υποχρεωτικών απαιτήσεων ήταν κάτι το ελάχιστο. Απλώς δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι τρία σημεία ήταν η παγίωση σε επίπεδο κράτους μέλους, τεχνική διαδικασία και συνέχιση αυτής της συζήτησης. Καταλήξαμε επίση στο ότι η ενδυνάμει αξία των συνόψεων αυτών βασίζεται σε δύο στοιχεία. Ανάλυση και ε, διασφάλιση εξοπιστίας. Αυτό όσον αφορά την προστιθέμενη αξία λοιπόν τον πρώτο χρόνο που είπαμε ότι είναι μάλλον χαμηλή. Θέλουμε επίσης να πούμε εδώ ότι τα ευρήματά μας ήταν ε, επίσης όσον αφορά την συμμόρφωση και όχι τόσο η αξία της ε, ετήσιας σύνοψης. Διαπιστώσαμε επίσης ότι τα περισσότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συνόψεις είναι περιτά, γιατί συμπεριλαμβάνονται σε άλλες εκθέσεις ή γιατί δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου σε εθνικό επίπεδο. Συστάσεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένες, με περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλουμε στο σημείο με αυτό για τις κατευθυντήριες γραμμές να υπάρχει μια εισαγωγή όσον αφορά την εθελοντική βάση. Οπότε θα θέλαμε να υπάρχει και κάποιο κίνητρο. Να υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που να δείχνουν την αξία του χειρήματος αυτού. Με κάποιο τρόπο να διατυπώνεται αυτό. Θέλουμε επίσης πρόσβαση του κοινού στις ετήσιες συνόψεις και στις δηλώσεις των κρατών μελών για τη διαχείριση. Τέλος θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε περισσότερο την το περιεχόμενο, την ποιότητα του περιεχόμενου και όχι μόνο της συμμόρφωσης. Μας ζητήθηκε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση και μας είπαν να επιταχύνουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πηδήξω μερικές διαφάνειες και να περάσω στα σημεία. Στα πιο σημαντικά σημεία της παρουσίασής μας. Λοιπόν, σχετικά με το, το, ε, σκέλος του ελέγχου ε, στην μελέτη μας Εάν δείτε την ε, διαφάνεια 28 θα δείτε ότι ουσιαστικά υπάρχουν ε, τρία βασικά θέματα για μας. Καταρχήν ε, η δήλωση της διοίκησης θα πρέπει να έχει επίσης ελεγχθεί ε, όσο αναφορά στοιχεία της από μια επαγγελματική εταιρεία οικονομικών ελεγκτών, ορκωτών λογιστών και ε, στη σελίδα 21 με 22 αναφέρουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης ε, και, ε, προσέγγισης και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θεωρούμε όμως ότι γενικώ ε, είναι μία ε, θετική προσέγγιση η οποία θα μπορέσει να συνδυάσει την ε, εθνική δήλωση ε, της διοίκησης ε, με την εργασία την οποία διεξάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή θα δούμε αν μία χώρα έχει ε, καλό ποιοτικό έλεγχο και πια όχι και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις συστάσεις μας, το οποίο δεν θα παρουσιάσω εκτενέως λόγω του περιορισμένου χρόνου. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει σημείο 6, πάμε στην απαλλαγή του 2007. Α, ορίστε. Έχετε κάτι να πείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες αυτής της μελέτης. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει υλικό προσκέψη κατά την απαλλαγή και θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα πρόγραμμα δράσης. Στη μελέτη αυτή έχουμε τις ετήσιες περιλήπτης οι οποίες έχουν περιορισμένη αξία και αν θέλουμε να προσθέσουμε και τις δηλώσεις της διοίκησης που υπάρχουν στο επόμενο παράρτημα ε, θα έλεγα ε, προς τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι καταρχήν μπορούμε να κάνουμε μία αξιολόγηση των ε, ετησίων περιλήψεων για το 2008 εφόσον στη μελέτη έχουν συμπεριληφθεί μόνο τα στοιχεία του 2007 και έχουμε μόνο προ εξαιρετικά τις ε, κινήσεις των κρατών μελών και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να υποφεληθούν από τα στοιχεία των άλλων ε, αλλά ε, θα περιοριστώ σε λίγα πράγματα γιατί τα επόμενα θα τα συζητήσουμε όταν θα έχουμε τις ακροάσεις των νέων επιτρόπων. Εδώ όμως ο Επίτροπος μας είπε ότι είναι πολύ προσιλωμένο σε αυτή την δήλωση της διοίκησης που του στηρίζει πολιτικά. Οπότε τι μέτρα έχουν ληφθεί συγκεκριμένα πέραν από αυτή την θετική αντιμετώπιση του Επιτρόπου και πότε μπορούμε να προσβλέψουμε προς αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριο Σοντίχτολο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο στόχος των ε, ετησίων περιλήψεων δεν είναι μόνο να δώσουμε οικονομικές πληροφορίες αλλά αποτελούν ε, ένα από τα στοιχεία μίας αλυσίδας οι οποίες πρέπει να γίνουν σεβαστές και ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο για να δοθεί μια θετική αξιολόγηση. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να φανεί σαφώς ότι το σύνολο του μηχανισμού αυτού ε, σέβεται τους διεθνείς κανόνες ε, οικονομικού ελέγχου και θα έπρεπε το θέμα αυτό να παραπευθεί στο ελεγκτικό συνέδριο για να μπορέσει να γνωμοδοτήσει σε αυτό το βασικό θέμα του προπολογισμού δηλαδή στο συσχετισμό μεταξύ ε, του απολογισμού και της θετικής δηλώσεως αλλά έχουμε ένα πολύ βαρύ μηχανισμό ελέγχου. Η ενδιάμεση, η ε, διοίκηση, οι ε, οικονομικοί ελεγκτές, όλοι αυτοί δεν μπορούν κάπως ε, να συμπεριλάβουν και έναν ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή διότι συμφωνώ σε αυτό θα έπρεπε λοιπόν να προσθέσουμε έναν εξωτερικό ελεγκτή για να δούμε ποια είναι το αποτέλεσμα και πώς αντιμετωπίζεται από τις εθνικές αρχές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημακάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και προηγουμένως ε, επένεσα τον κύριο Κάλλας διότι έκανε ε, την συνόψη αυτή και ε, μας την παρουσίασε. Πρέπει όμως να σας πω ότι το αποτέλεσμα είναι περιορισμένο. Συμφωνώ δηλαδή με την κυρία Ντελάνιε. Το ερώτημά μου είναι το εξής ε, τι έχουμε ακόμη μπροστά μας, ποια οδό έχουμε ακόμη να διανύσουμε διότι αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να πιέσουμε ε, για τις εθνικές δηλώσεις αξιοπλησίας και δεν θα πρέπει εδώ να πρόκειται απλώς για ένα εικονικό φάρμακο ε, ενοχλούμε πρέπει να σας πω διότι ατυχώς δεν έχουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα δεν έχουμε δηλαδή δηλαδή την αξιοπιστία την οποία επιζητούμε. Πού βρισκόμαστε στο 10-15% ή κάτω και από αυτό το επίπεδο. Ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εσείς εδώ παρουσιάσατε το πρώτο πόσα τις συστάσεις σας. Μπορείτε να μας πείτε αν ε, υπολογίσατε πόσο θα κοστίσει η εφαρμογή του συστήματος αυτός άμεσα, έμεσα και συνολικά. Διότι θα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα, ε, θα πρέπει να προβλέψουμε και εκπαίδευση. Όλα αυτά μαζί τι θα κοστίσουν. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Όταν τα βλέπουμε, όντως μπορούμε να πάθουμε παράνοια, διότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ μακριά και επανερχόμεθα σε αυτό το οποίο ακούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, ένα μέλος ε, του κοινοβουλίου του προπολογισμού της κοινότητος ε, αποδίδεται χωρίς σχόλιο και είναι εξωτερική βοήθεια. Και ε, μετά ε, χρειάζεται δημοσιονομικά η κοινότητα τη συνδρομή των κρατών μελών. Τι γίνεται λοιπόν με την αξιοπιστία. Πρέπει να βρούμε μια εύκολη λύση και όχι δύσκολα και περίπλοκα θέματα. Ο κ. Κάλλα έφυγε. Υπάρχει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να δώσει κάποιε απαντήσει όσα μα είπαν οι βουλευτέ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο Αντιπρόεδρος, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή η μελέτη πρέπει να εξεταστεί μέσα στο σωστό πλαίσιο. Είναι ε, για τον πρώτο χρόνο, δηλαδή για το 2007. Δηλαδή ήδη το 2008 έχουμε σημαντικές βελτιώσεις, δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη έχουν καλύψει τις ε, ελάχιστες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 7 από τα νέα κράτη έχουν έχουν συμμορφωθεί στην πρόσκληση η οποία έγινε στις κατευθυντήριες γραμμές και έχουν ε, επισυνάψει στην ετήσια έκθεση μία δήλωση διαχειριστική ε, όπως ελέγχθη. Δεν πρέπει λοιπόν να απογοητευόμαστε. Υπάρχουν θετικά στοιχεία και η μελέτη αυτή μας δείχνει μεθοδολογικά τι πρόοδος μπορεί να γίνει και προσπαθούμε απλούστατα. Η κυρία Ντελάνια περιμένει την απάντησή μου και θα ήθελα να σας πω ότι τις εθνικές δηλώσεις δεν τις θέλει το Συμβούλιο και το λέει ρητός. Οπότε εμείς συνεργαζόμαστε ε, οικειοθελώς με τα κράτη-μέλη που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Και βεβαίως δεν ε, ε, χρονοτριβούμε και έχουμε πει ποιο είναι το ελάχιστο θέμα με το οποίο θα προχωρήσουμε βάσει των στοιχείων διότι κάποιος είπε ήδη ότι έχουμε τις συνδρομές των κατών μελών αλλά είναι τελείως διαφορετικές οι παρουσιάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο το οποίο θα μας βοηθήσει στην αξιολόγηση. Όσο αναφορά τις ε, οικειοθελείς ε, ε, δηλώσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο με αλλαγή νομική. Υπάρχει τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία υπάρχει επισήμως συναπόφαση του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο και θα υπάρχουν ε, εξελίξεις αλλά αντιλαμβάνεστε τη θέση μου θα υπάρξει μια νέα επιτροπή και μετά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε απλώς σχολιάζω τα ερωτήματα τα οποία μου ετέθησαν τουλάχιστον στον κύριο Οντή θα ήθελα να το υπενθυμίσω ότι οι αιτήσιες ε, οι δηλώσεις ε, είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας όπου παρεμβαίνει και η δήλωση εξοπιστίας. Αλλά χρειαζόμαστε ε, μεθοδολογικά μία σωστή οδό και βεβαίως το ελεκτικό συνέδριο θα προσέξει πάρα πολύ τη μεθοδολογία που θα υιοθετηθεί. Το αντιλαμβάνομαστε, ξέρουμε ότι ε, θα πρέπει ε, όλοι να συμφωνήσουν στη μεθοδολογία αυτή. Ξέρετε λοιπόν πώς πόσο ανεξάρτητα είναι ορισμένα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και ιδίω τη χώρα από την οποία προέρχεστε κύριε Οντή. Οπότε δεν ξέρω αν θέλετε απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις, αλλά έχουμε και συναδέλφους από τα διαρθρωτικά ταμεία για να απαντήσουν σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κνέντλερ έχει το λόγο αν θέλει να απαντήσει στον κύριο Οντί Λιμπερντάτσκι και στους άλλους που πήραν τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρώτο θέμα, το πρώτο ερώτημα αναφερόταν στον υπερβολικό έλεγχο. Αν κοιτάξετε προσεκτικά την εικόνα θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα ελέγχων. Τώρα, αν κάποια από τα επίπεδα μπορεί να εγκατελειφθεί ή όχι, δεν μπορώ να απαντήσω τόσο εύκολα. Απ' την άλλη, αναφερθήκατε και στις ευθύνες προδιαγραφές ελέγχου. Πρέπει να βασιστούμε σε κάποια... Ο βασικός ελεγκτής πρέπει να βασίζεται στο έργο που έχει κάνει άλλος ελεγκτής. Μπορεί να το κάνει αυτό. Αν το κάνεις αυτό μπορεί να αποφύγεις ε, επικαλύψεις προσπαθειών. Δεν χρειάζεται να εξαλειφθούν κάποια από τα επίπεδα. διότι περιπλέκονται τα θέματα σε εθνικό επίπεδο, σε συνταγματικούς τομείς και δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ θα προτιμούσα να ακολουθούμε τη μέθοδο του να βασιζόμαστε σε έργο άλλων ελεγκτών αντί να αφαιρούμε επίπεδα ελέγχων. Και κυρίως να μην σε θέματα που αφορούν σε εθνικό επίπεδο ελέγχους που απορρέουν από τα εθνικά συντάγματα. Τώρα, το, το αποτέλεσμα πλασίμπο που αναφέρθηκε. Στη μελέτη μας είδαμε ότι υπάρχουν κάποια ωφέλη, μικρά ωφέλη από τις ετήσιες εκθέσεις. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι ετήσιες εκθέσεις, οι συνοπτικές, είναι χρήσιμες μόνο αν συμπεριφθούν στην εθνική δήλωση. Απλώς, απλώς παρουσιάζουν στοιχεία. το κόστος του συστήματος. Θα είμαι ειλικρινής. Δεν κάναμε υπολογισμό κόστους. Δεν τόσο δαπανηρό όμως, διότι υπάρχουν οι θεσμοί. Αυτό που χρειάζεται είναι να συναθρήσεις κάποια στοιχεία και να εφαρμόσεις κάποια συστήματα. Δεν χρειάζεται δημιουργία κάποιου φορέα. Χρειάζεται καλύτερο σύστημα. Να είσαι πιο συστηματικός. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις κάτι. Χρειάζεται αναδιάρθρωση φυσταμένων συστημάτων. Και πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ δαπανηρό. Άλλο ερώτημα. Άλλα μέσα. Άλλους τρόπους αντί δήλωση αξιοπιστίας ή μάλλον εθνικές δηλώσεις διαχείρισης. Πιστεύουμε ότι καμιά φορά η έμπνευση για το δημόσιο τομέα μπορεί να προέρχεται από τον ιδιωτικό. Σχετικά με αυτό, χρήσιμα είναι αυτά που ήδη θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα φυστάμενα Υπάρχουν κάποιες εθνικές πρωτοβουλίες για την εισαγωγή μέσων, εργαλείων για εθνικούς προϋπολογισμούς, όχι μόνο για πόρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και για εθνικούς προϋπολογισμούς. και αυτά τα μέσα επηρεάζουν το ένα το άλλο αν θέλετε. Τα αποτελέσματα του ενός επηρεάζουν το άλλο. Τέλος, δεν πιστεύουμε ότι οι εθνικές δηλώσεις είναι η πανάκια για, το εν μέρη, για την εν μέρη αρνητική δήλωση εξοπιστίας. Δεν είναι απλά τα πράγματα βέβαια. Αλλά αν εφαρμόσουμε εθνικές δηλώσεις διαχείρισης. Αυτό θα επηρεάσει άμεσα τα συστήματα, τα εθνικά ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου. Και έτσι θα μειωθεί το επίπεδο των σφαλμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Στον κύριο Εγκβίρδα δίνω το λόγο, μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο εδώ να πούμε πως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όπως είπε και ο κύριος ε, Ταβέρν, ότι η συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα είναι ζήτημα κυρίως μεθοδολογίας και γι' αυτό οι συνάδελφοί μου στο Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν αρχίσει συζητήσεις με τρία εθνικά ελεγκτικά όργανα των κάτω χωρών της Δανίας και της Τσεχίας προκειμένου να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε κοινού ελέγχους μαζί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με τα εθνικά όργανα ελέγχου των τριών αυτών χωρών. Είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα. Να δούμε, θα είναι κοινή έλεγχη, συντονισμένη έλεγχη, θα δούμε, ώστε ε, να περιοριστούν και οι δαπάνες. Καλό θα ήταν αυτό να είναι γνωστό. Ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις τους. Ορίστε. Ο κύριος Εουντή. Ευχαριστώ πολύ σύντομα για αυτό το θέμα που βέβαια και έχω στην καρδιά μου. Είπατε μεθοδολογία. Η μεθοδολογία διακανονίζεται περίπου από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα διεθνή πρότυπα ελέγχων που εφαρμόζουν όλοι όταν πρόκειται σε διεθνές επίπεδο ελέγχους. Οπότε η μεθοδολογία, η κοινή μεθοδολογία υπάρχει. Τώρα αν το ελεγκτικό συνέδριο, το γαλλικό, αρνείται, είναι για δύο λόγους. Πρώτον, τη απουσία νομικής βάσης δεν θέλει να είναι κάτω από το Ευρωπαϊκό Ολεκτικό Συνέδριο και δεύτερον οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι πάρα πολύ λίγοι στο σύνολο των κονδυλίων που έχει το κράτος μέλος. Τώρα έχουμε τη Λισαβόνα με μια νομική βάση και η οποία επιτρέπει, και καλό θα ήταν να ξέρουμε τι λέει γι' αυτό το Ολεκτικό συνέδριο, νομική βάση λοιπόν που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Ολεκτικό Συνέδριο να ζητήσει από οποιαδήποτε δίκηση που έχει ελεκτικές ε, αρμοδιότητες, προκειμένου δηλαδή να δώσει ΝΤΑΣ, να ζητήσει λοιπόν συνεργασία. Αυτή η νέα νομική βάση είναι πολύ βασική και αλλάζει την έννοια της συνεργασίας έτσι όπως την ξέραμε από τις προηγούμενες συνθήκε. Ευχαριστώ. Απαλλαγή 2007, το σημείο 7 της ημερήσιας διατάξης. Δίνω το λόγο στον εισηγητή Σόντεργαρντ. <clears throat> Øh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ με, μια, ε, με τις ευχαριστήσεις μου για όλους σχετικά με ε, την συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συντονιστές και τους κοιόδης εισηγητές και τη γραμματεία που έκανε εξαιρετική δουλειά και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω την κυρία Σεν για την συμμετοχή της παρόλο που η πολιτική της ομάδα κατέληξε στις αντίθετες, στα αντίθετα συμπεράσματα από ε, τα δικά μου. Η κυρία Αντρέα Σεν και η ομάδα της μας λέγει να απορρίψουμε την τροπολογία 14 ενώ εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται εφόσον έχουμε παραχωρήσεις από το Συμβούλιο, παραχωρήσεις τις οποίες δεν είχαμε επιτύχει ποτέ στο παρελθόν και αυτές τις ε, παραχωρήσεις πρέπει να τις αξιοποιήσουμε για την μελλοντική μας σχέση με το Συμβούλιο σχετικά με τις απαλλαγές γιατί προχωρήσαμε πολύ. Πριν από ένα χρόνο το Συμβούλιο, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου μάλλον είχαν βγει από τη συνεδρίαση, είχαν εγκαταλείψει τη συνεδρίαση όταν μιλήσαμε για την αιτήσια απαλλαγή τους. Και στο παρελθόν το Συμβούλιο έχει αρνηθεί να απαντήσει στις γραπτές μας ερωτήσεις. Και στις 26 Σεπτεμβρίου ήταν η τελευταία φορά που μας προσκάλεσε το Συμβούλιο να συμμετάσχουμε σε ένα άτυπο γεύμα ε, το μεσημέρι για να συζητήσουμε τις ετήσιες απαλλαγές αλλά αυτά έχουν αλλάξει τώρα άλλαξε η κατάσταση γιατί καταρχήν έχουμε πραγματικές συναντήσεις με το Συμβούλιο και ε, παίρνουμε και μία σαφή απάντηση ή στις γραπτές μας ερωτήσεις. Βέβαια δεν είναι όλα τέλεια και πολλές από τις απαντήσεις είναι είτε λαθασμένες, είτε ε, ε, ελλειπείς. Και ε, ε, το Συμβούλιο επιμένει να, οι συναντήσεις να είναι άτυπες ακόμη και αν έχει μεταφραστές, ε, γραμματεία, συντονιστές και πρακτικά της συνεδρίασης. Αυτό όμως το οποίο πετύχαμε είναι ότι απάντησαν στις ερωτήσεις μας και μπορούμε να συναντηθούμε με το Συμβούλιο επίσημα με διερμηνείς ακόμη και αν το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι άτυπη συνάντηση και αυτό πρέπει να αποτελέσει την βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις για την απαλλαγή του Συμβουλίου και αυτό είναι το περιεχόμενο της προτάσεως το οποίο υπάρχει τώρα και ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσει να υιοθετηθεί. Δεν θέλω βέβαια να υπερβάλλω αλλά πρέπει να σας πω ότι προς παρόν έχουμε κερδίσει μία μάχη αλλά όχι τον πόλεμο για τη διαφάνεια και την ε, ε, σαφήνεια. Αν ε, λοιπόν θέλουμε να καταλήξουμε θα χρειαστεί εγκαίρως να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο. Δεν πρέπει δηλαδή να περιμένουμε, θα πρέπει από την αρχή το Συμβούλιο να συναντιέται μαζί μας, να μας δίνει καλύτερες τις απαντήσεις, να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε τις απαντήσεις του και να ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις. Αλλά στο μέλλον οι συζητήσεις θα είναι σε υψηλότερο επίπεδο και ελπίζω ότι θα υπάρξει στήριξη για τις προτάσεις τις οποίες διατυπώνουμε, ιδίω όσον αφορά τις ε, τροπολογίες επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει. Διότι υπάρχει μία ενιαία γνώμη, έχουμε δύο προφορικές ε, ε, συμβιβαστικές προτάσεις οι οποίες αντικαθιστούν 7 τροπολογίες και έτσι υπάρχει μία πιο ομοιόμορφη ε, παρουσίαση υπάρχουν και προφορικές τροπολογίες και πέντε πολιτικές ομάδες μας στηρίζουν άρα υπάρχει σαφή στήριξη σχετικά με τις δύο προφορικές τροπολογίες οι οποίες υπάρχουν είναι μια καλή σύνοψη των προτάσεων τις οποίες ε, θέλουν να ε, αντικαταστήσουν και είναι όπως είπα συμβιβαστικές και μπορούμε να τις στηρίξουμε και τις δύο. Όσον αφορά την διατύπωση, ίσως ε, δεν είναι πάντοτε σε όλα τα σημεία σαφής και ελπίζω οι συνάδελφοι να προτείνουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η διατύπωση. Ε, ε, υπάρχει μία προσθήκη στην πρώτη συμβιβαστική τροπολογία για αλλαγή ορισμένων όρων και θα έλεγα να τη στηρίξουμε. Όσον αφορά την πρώτη ε, τροπολογία την έχω αγγλικά και λέγει ότι εις την διαθεσμική συμφωνία αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα παράρτημα σχετικά με την δημοσιονομική διαδικασία απαλλαγής. Οι πρώτες ε, λέξεις θα πρέπει να αλλάξουν αντί ε, για encourages να πούμε ε, ε, απαιτεί ε, να υπάρξουν. Και με τις παρατηρήσεις αυτές θέλω τώρα να ανοίξω τη συζήτηση και ελπίζω ότι αύριο στην ψηφοφορία θα υπάρξει ευρεία στήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πραγματικά, ευχαριστώ όλους για τη δουλειά αυτή που έγινε, που ήταν πολύ περίπλοκη, αλλά μας επιτρέπει να σημειώσουμε πρόοδο, κυρίως όσον αφορά τη θεσμική αξιοπιστία, πολύ σημαντικά βήματα σε όλο το Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας ειδικά. Υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει όσον αφορά το σημείο αυτό. Κανένας. Ορίστε, κύριο Ντί. Ναι, να πω μία λέξη όσον αφορά την τροπολογία μου 5, όπου είδα κύριε Σιγητά ότι προτείνατε αρνητική ψηφοφορία και νομίζω ότι και άλλοι θα έχουν αντίρρηση όσον αφορά αυτή την τροπολογία. Προτείνει να μελετήσουμε τη νομική βάση βάση της οποίας η Επιτροπή μας δύναται ή δεν δύναται να εργαστεί όσον αφορά τις δαπάνες και τις οικονομικές συναλλαγές του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιχειρήσεις στατιωτικές και την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Διστάζω σε αυτή την τροπολογία, διότι βλέπω ότι στο συμβιβασμό προτείνεται να υπάρχουν διοργανικές συμφωνίες. Αναγνωρίζετε δηλαδή ο ίδιος ότι υπάρχει ένα νομικό, νομική θεά ζώνη εδώ. Και είδα και διαφοροποίηση από την πρώτη έκθεση μέχρι τόσο από τη στάση σας. Λυπάμαι. Διότι δεν υπάρχει αυτή η μελέτη. Διότι όσον αφορά τη σχέση με το Συμβούλιο, που ξεκινά η συνεργασία τη συνθήκη τη Λισαβόνα, προβλέπονται άλλα. Βλέπετε τι προβλήματα έχουμε με την έκθεση Μπροκ και του αρχηγού ε, κρατών κυβερνήσεων αφορά τι εξωτερικέ υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Θα είναι δικυβερνητική η φύση του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να ελέγχει. Οι πολιτικέ διαπραγματεύσει μόλι τώρα αρχίζουν. Εγώ θα ζητούσα να διεξαχθεί μια μελέτη. Να ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μα. Δεν είμαι σίγουρο ότι τα γνωρίζουμε και στο θέμα αυτό του Συμβουλίου εγώ έχω το συνέστημα ότι μένει κάτι ατελείωτο. Δηλαδή θέλω να ξέρω ποια είναι τα δικαιώματα της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να διεξαχθεί η μελέτη όπως είπα και πριν. Λυπούμε που βάλατε αρνητικό πρόσημο στην τροπολογία μου. Ευχαριστώ. Αμερχάουζερ. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα το όνομά μου έτσι όπως το προφέρατε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την έκθεση σχετικά με την απαλλαγή του Συμβουλίου διότι απεδείχθη ότι πολλά ε, από τα ερωτήματα που είχαμε θέσει παραδείγματο χάρη στο σημείο 22α ή δεν έχουν απαντηθεί καθόλου ή ανεπαρκώς και υπάρχουν απαιτήσει που διατυπώσαμε στο πρώτο σχέδιο εκθέσεως ε, ότι είχαμε πει ότι δεν ήταν πλήρες τώρα βλέπουμε ότι κανένας λογαριασμός δεν έχει κλείσει και δεν ξέρουμε καν αν το Συμβούλιο ε, προτίθεται να κλείσει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς. Όταν λέμε λοιπόν ότι παρακαλούμε το Συμβούλιο να μας στείλει ε, ένα μια ετήσια έκθεση ε, διοικήσεως ε, είναι ε, προφανές ότι εμείς είμαστε οι ελεγκτές και δεν πρέπει να πηγαίνουμε παρακαλετά Στην ε, προηγούμενη Ολομέλεια είχαμε πει ότι απαιτούμε ε, να έρχονται όλα τα θέματα εις ε, την δημοσιονομική αρχή του, του Κοινοβουλίου και δεν μπορούμε να μιλάμε για το Συμβούλιο για απόδοση λογαριασμών και δεν νομίζω ότι μπορούμε μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε με την απαλλαγή αυτή και για τους λόγους που προανέφερα δεν θα την υπερψηφίσω. Η κυρία Ανδρέασεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο με τον συνάδελφο. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του. Δεν πήραμε απάντηση σε καμία ερώτηση μας. Εδώ εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και είμαστε εδώ για να εγκρίνουμε την ε, σωστή διαχείριση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν πήραμε τις αναγκαίες απαντήσεις, άρα δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Διαρωτώ με. Είμαι περίεργος. Ποια είναι η συμπεριφορά της Επιτροπής, διότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο περιόρισε τα σχόλιά του στα λογιστικά του Συμβουλίου σε 30 γραμμές. Και αυτή η Επιτροπή αποφάσισε να διεξάγει έρευνα. Και δεν είναι στα καθήκοντα της Επιτροπής η διεξαγωγή έρευνας. Ποιος ο σκοπός διεξαγωγής της έρευνας που έπρεπε να έχει διεξαχθεί το ελεκτικό συνέδριο και απλώς έτσι να καταργήσουμε τα όρια και να χορηγήσουμε απαλλαγή. Αφού θέσαμε ερωτήσει και δεν πήραμε απαντήσει. γιατί αποφασίζουμε πολιτικά ότι θα δώσουμε απαλλαγή και να διαγράψουμε την παράγραφο που εκφράζουμε ανησυχίε όσον αφορά τα λογιστικά του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την, ε, τον εισηγητή ε, για την έκθεση και πιστεύω ότι έχουμε προχωρήσει. Έχουμε επιτύχει περισσότερα από όσα περιμέναμε. Πιστεύω ότι όλες οι συμβαστικές προτάσεις είναι καλές και θα τις στηρίξω. Θα ήθελα να πω στον συνάδελφο Όντι ότι είναι καλή ιδέα να γίνει αυτή η μελέτη ουσιαστικά και του υπενθυμίζω τη συζήτηση που είχαμε με το Συμβούλιο και με την Γραμματεία του Συμβουλίου όπου μας δόθησαν διάφορες ερμηνείες ιδίως από, από έναν Γάλλο εκπρόσωπο του Συμβουλίου που είναι πολύ έξυπνες. Δεν θεωρώ ότι εάν προβούμε σε μία μελέτη θα προχωρήσουμε. Πολιτικά έχουμε ήδη προχωρήσει και αυτή η πολύ αργή πορεία πρέπει να συνεχιστεί και ίσως μπορέσουμε να αλλάξουμε τη διαδικασία. Έχω να κάνω μία ερώτηση στην κυρία Γκρέσλε και στον εισηγητή σχετικά με την τροπολογία 4 για το ποιες επιτροπές είναι αρμόδιες ε, διότι ο εισηγητής μιλάει για μία επιτροπή η κυρία Γκρέσλε για πολλές επιτροπές μπορείτε να μας τις ονοματίσετε υποθέτω ότι είναι η κομπού και η κοκομπού δηλαδή η Επιτροπή Προπολογισμού και Ελέγχου Προπολογισμού αλλά αν γράψουμε ρητός τι εννοούμε νομίζω ότι θα αποφύγουμε τη παρανοήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Ζόντερκαρτ για την έκθεσή του διότι μετά από μακρές και επίπονες συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα έχει επιτύχει ένα αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είναι πολιτική επιτυχία ότι είχαμε μία συζήτηση με το Συμβούλιο. Έχω κατανόηση για τις επιφυλάξεις της κυρίας Ανδρέας και του κυρίου Έρενχάουζερ αλλά σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε ευγνώμενοι όταν μας παίρνουν στα σοβαρά σαν συνομιλητές και απαντούν στις ερωτήσεις μας. βέβαια ίσως αυτή είναι αντιμετώπιση ενός νέου ευρωβουλευτή ε, ο οποίος δεν έχει μακρά πείρα ε, ιδίως όταν βλέπουμε πως το κοινοβούλιο ε, ποιας μεταχείρισης μάλλον την χάνει το Κοινοβούλιο από τα κράτη-μέλη και είναι ακόμη πιο αξιοπερίεργο να συνυπολογίσουμε ότι για τη δουλειά μας υπάρχουν πολύ σαφές, σαφείς διαδικασίες οι οποίες βασίζονται σε μια συμφωνία κυρίων της δεκαετίας του 70 Οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα που επιτύχαμε και συμφωνώ πλήρως με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Χατζημαρκάκης. Έχουμε ανοίξει μία πολιτική οδό όπου απαιτούμε όσον αφορά τις διαδιαδικασίες να υπάρχουν σαφές σχέσεις και σαφές ευθύνες και επ' αυτής της βάσεως παρόλο που ε, με απογοντεύει ο αριθμός ε, των ε, θεμάτων που έχουν να μείνει ακόμη σε εκκρεμότητα να αξιολογήσω διαφορετικά από την κυρία Αντρέσεν και τον κύριο Χάουζερ το αποτέλεσμα. ναι, τα οποία είναι ανοιχτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε τώρα να τα διευκρινίσουμε αμέσως διότι τότε θα λέγαμε ότι δεν μπορούμε να προβούμε στην απαλλαγή αλλά το Συμβούλιο ακολουθεί ακολουθεί το δρόμο του θα συνεχίσει στα θέματα αυτά και τουλάχιστον αυτό είχαμε συμφωνήσει στη συνεδρίαση των συντονιστών ότι το Κοινοβούλιο θα εμείνει στα θέματα αυτά και θα απαιτήσει διευκρινήσεις. Δεν υποχωρούμε δηλαδή αλλά όπως το είπε και πολύ, ο, πολύ ωραίο κύριος Σόντερ Γκάρντεν, δεν υποχωρούμε μεν, συνεχίζουμε να μαχόμαστε, αλλά θα θέλαμε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή τη διαθεσμική συμφωνία και να πετύχουμε ε, και να πετύχουμε. Οπότε, ε, εάν ε, θεωρήσουμε αν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο, θα λέγαμε ότι είναι μισογεμάτο και μπορούμε να προχωρήσουμε. Κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, ε, τιμιότητα και το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο ε, προχωρήσαμε και διαπραγματευτήκαμε τα θέματα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι ο προπολογισμό του Συμβουλίου είναι μία μαύρη τρύπα, δεν ξέρουμε πού πάνε τα χρήματα και οι γενικές γραμμές είναι γνωστές. Και αυτό που πάντοτε μας ενοχλούσε ήταν η η χρήση των ε, ε, τακτικών ε, δημοσιονομικών μέσων στην εξωτερική πολιτική. Βέβαια όμως όλα αυτά δεν αποτελούν αιτία να αρνηθούμε την απολογή. Βεβαίως ορισμένοι είναι πιο ριζικοί αλλά μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις και εγώ είμαι ικανοποιημένη με τη θέση μου. Θα ήθελα να πω στον κύριο Ντί ότι χάρη εις την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας επιτέλους η κατάσταση αλλάζει ε, και ελπίζω ότι σε δύο χρόνια θα μας ενδιαφέρει ε, και εμάς η μελέτη αυτή οπότε Ζων Πιέρ νομίζω ότι θα είναι καλό καλό είναι να γνωρίζουμε βάσει ποιας νομικής βάσεως λειτουργούμε και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή αλλά θα έπρεπε να πω ότι ε, δεν χρειάζεται να διατηρήσουμε περαιτέρω μία μεσαιωνική ε, δομή η οποία υπάρχει όπου ένα ελεύθερα εκλεγμένο κοινοβούλιο θεωρείται υποτακτικό στο Συμβούλιο. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τέτοιες μεθόδους στον 21ο αιώνα και γι' αυτό θεωρούμε ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να επιζητήσει από κοινού με εμάς να βρει λύσεις και πιστεύω ότι στην διαθεσμική συμφωνία θα τις ε, επιζητήσουμε και θα τις ε, ε, βρούμε και πιστεύω ότι δεν πρέπει να αρνηθούμε την απαλλαγή αρκεί να ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε ε, και αυτό μας οδηγεί σε μια τελείως διαφορετική άποψη από ό,τι είχαμε προκαιρού. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους διότι θέλουμε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι πρόκειται για μια κοινή για ένα κοινό μέλημα του Κοινοβουλίου και γι' αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ριβελίνη, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι παράξενο ότι τη στιγμή που ότι λέμε ότι είναι αρχή μιας μάχης, μιας συζήτησης, όπως είπε συνάδελφος, ότι ξεκινάει μια μάχη, μετά κάποιος να έχει αντίρρηση όσον αφορά την εμβάθυνση όπως ζητά ο συνάδελφος Οντί με την τροπολογία του. Δηλαδή κατά τρόπο κατανοούμε τελικά ποια είναι τα όρια της μάχης. Και προσπαθούμε να κάνουμε μια μάχη αλλά δεν ξέρουμε με ποια πυρομαχικά μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη μάχη. Συμφωνώ ότι είναι σωστό ίσως να περιμένουμε τη Λισαβόνα αλλά μετά να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι τα όρια, τα όρια των δράσεων μας, των δράσεων του Συμβουλίου θα ήταν κάτι καλό. Εγώ θα υπερψηφίσω λοιπόν την τροπολογία του συναδέλφου του κυρίου Οντί, θα υπερψηφίσω και περιμένοντας ίσως και τη συνθήκη της Αβώνας και μετά κάνουμε δελεχές στη συζήτηση διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρουμε τα όρια μας, για να ξέρουμε ε, ποιες θα είναι οι δράσεις που θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Σόντεργαρντ, κύριε Σόντεργαρντ, θέλετε να απαντήσετε σε αυτά ερωτήματα του κυρίου Χατζημαρκάκη και την ε, και όσα υπόθηκαν γύρω από την ε, τροπολογία. Απάντηση του κυρίου Σόντερμαρκ. Όσον αφορά αυτή την πρόταση, αυτή την τροπολογία, πρέπει να πω ότι οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται ότι οι οι άλλε επιτροπέ που ενδιαφέρονται είναι η ΑΦΕΤ, η Επιτροπή Προπολογισμών επίση, εκτό από τη δική μα επιτροπή. Είναι ένα θέμα επίση εξωτερικών υποθέσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για κονδύλι που προβλέπεται για την ασφάλεια και την άμυνα. Θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Αυτό τίθεται σαν ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Δεν υπάρχει τροπολογία. Εμένα με ικανοποιεί αν είναι κάπως αόριστη διατύπωση. Αλλά δεν έχω και κανένα πρόβλημα για αντίθετη πρόταση. Μια συγκεκριμένη αναφορά στην Επιτροπή που αναφέρατε. Κύριε Οντί, θα ήθελα να πω ότι δεν τίθεται το θέμα αν είναι καλή ιδέα η έρευνα ή όχι. Θέλουμε να ξέρουμε αν ναι ή όχι, εδώ είναι ο σωστός χώρος για να ζητήσουμε τέτοια έρευνα. Αν είναι η καλή στιγμή. Εγώ νομίζω ότι ίσως δεν είναι η καλύτερη χρονική στιγμή θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ενδεχομένως τη νομική υπηρεσία να μας κάνει κάποια ε, πρόταση, κάποια διευκρίνηση νομική υπηρεσία και μετά συζητάμε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα αυτό. Εγώ δεν, δεν κρίνω την ιδέα σας αν είναι καλό να πούμε ναι ή όχι σε μια έρευνα. Δεν ξέρω αν είναι ο χώρος σωστός και η ώρα σωστή. Τώρα, όσον αφορά τις διάφορες επικρίσεις που ακούστηκαν, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν βρήκαν απάντηση. Ναι, το είπα ο ίδιος στην αρχή. Πράγματι, ισχύει αυτό. Αν αναφερθήκατε σε κάτι, αναφέρατε κάποια παραδείγματα, με αναφερθήκατε σε πιστόλι, σε όπλο κλπ. για να, πάρετε, να προβάλλετε την εικόνα του πολεμιστή που πρέπει να έχουμε. Εάν υιοθετηθεί αυτή η τοποθέτηση από την πλευρά της Επιτροπής μας, θα πρέπει να καθορίσουμε κάποιους αφέστατου προσανατολισμούς που θα αποτελέσουν αφετηρία των μελλοντικών στρατιών. Μετά μπορούμε να δούμε αν θα πετύχουμε πρόοδο ή όχι. Βλέποντα και κάνοντα, Όταν διορίστηκα εισηγητή, εξέτασα όλα τα ψηφίσματα που είχαν ε, περάσει τα τελευταία χρόνια και διαπίστωσα ότι σε κάθε ψήφισμα, σχεδόν σε κάθε ψήφισμα, διαμαρτυρόμαστε, λέγαμε, δεν πήραμε απάντηση, δεν έγινε συνάντηση, δεν έγινε συνεδρίαση κλπ. κλπ. Αν αρνηθούμε σήμερα θα γίνουν τα ίδια του χρόνου και του παραχρόνου. Σήμερα έχουμε μια λύση, κάναμε μια διαπίστωση και λέμε κάποια πράγματα. Λέμε ότι πρέπει να επιβάλλουμε συνεδριάσεις στο Συμβούλιο υπό τη μορφή αυτών των συναντήσεων. Είναι μια φετηρία. Ε, και νομίζω ότι είναι μία πρόοδος. Βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο μακριά, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Το πιο εύκολο βέβαια είναι να ζητήσουμε περισσότερα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της πλειοψηφίας. Πρέπει να έχουμε πλειοψηφία που θα υποστηρίζει το κείμενο. Νομίζω ότι είναι εφικτό, είναι μια καλή ευκαιρία. Βέβαια κάποιοι λένε πρέπει να προχωρήσουμε πιο μακριά κλπ αλλά πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή αφετηρία. Και πολλά θέματα εκκρεμούν, πράγματι. Ισχύει. Και στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις. Σύντομα, μάλιστα, θα συναντήσουμε σε κάποιες εβδομάδες ε, τους διάφορους αρμοδίους. Πράγματι, ίσως Ίσως να κρατάμε νεροπίστολο και να βγαίνει έτσι ένα πίδακας νερού από ένα νεροπίστολο αυτή η πρόοδο μα, αλλά παρόλα αυτά ε, είναι μια προσπάθεια. Ευχαριστώ. Αντρέασεν. Κυρία Αντρέασεν. Νομίζω ότι ο μόνος προσανατολισμό που έχουμε καθορίσει με το όλο εγχείρημα είναι ότι θα δεχθούμε ανοησίε στο μέλλον σαν απάντηση όπως κάναμε και σήμερα. Καλώς, ευχαριστώ. Έχουμε και άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη και έχουμε μόλι ένα τέταρτο. Λοιπόν, γι' αυτό αν δεν έχετε άλλε παρεμβάσει, σα προχωρήσουμε. Σημείο 8. Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την σχεδίου τη Επιτροπή στον Τομέα τη Δικαιοσύνη των Εσωτερικών Υποθέσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, κύριο Ολμπριχτ. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις όσον αφορά το θέμα μας αυτό. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για την έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. 2000 με 2006, μάλλον 2001 διορθώνω μιλητής 2006. Πρόκειται δηλαδή για αξιολόγηση δραστηριοτήτων. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε τις δραστηριότητες της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο όπως είχε γίνει σε άλλες περιπτώσεις τις διαδικασίες αλλά και τα συγκεκριμένα γεγονότα επιτόπου. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε στην έκθεση ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Όμως γενικά μιλώντας αυτό που προσπαθώ να βάλω εγώ στην έκθεσή μου είναι πρώτα απ' όλα ότι σημειώνουμε πως πρόκειται γενικά για μια θετική γνωμοδότηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως γενική παρατήρηση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική γενικά, δηλαδή δίνει μια σχετικά θετική αξιολόγηση του ελεγκτικό συνέδριο. Στη συνέχεια η έκθεση αυτή δείχνει ότι τέτοιου είδους πολιτική πρέπει να συνεχιστεί. Με διαφορετικούς τρόπους. Επίσης όμως είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι το λεκτικό συνέδριο στην έκθεσή του δείχνει τα διάφορα είδη αποτελεσμάτων που έχουμε, διαφορετικής ποιότητας δηλαδή. Η ποιότητα των λεγόμενων προγραμμάτων επενδύσεων, η απόδοσή τους, η βιωσιμότητά τους είναι μεγαλύτερη από ότι η προσπάθεια οικοδόμησης θεσμών στις χώρες αυτές. Εκεί σημειώνονται δυναμίες. Γι' αυτό εξάλλου στην έκθεση αυτή μπορούμε να διαβάσουμε ότι χρειάζονται και άλλες δραστηριότητες για να υπάρξει μεγαλύτερη σύνδεση ανάμεσα στις επενδύσεις και την ε, βιωσιμότητα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, πιστεύω, που βρίσκουμε στην έκθεση αυτή. Κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον στην έκθεση αυτή του λεκτικού συνεδρίου και το περιλαμβάνω και εγώ στη δικιά μου έκθεση είναι η έκκληση που γίνεται προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει ό,τι μπορεί παραπάνω για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δωρητών επιτόπου. Γιατί βλέπετε και αυτό είναι ένα σημείο αδυναμίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο δωρητή, αλλά πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δωρητών. Τώρα για να συνοψίσω, Πρόεδρε, πιστεύω ότι διαβάζοντας την έκθεση αυτή του λεκτικού συνεδρίου, πρώτον, πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια θετική αξιολόγηση, όχι μόνο επί των διαδικασιών, αλλά και επί των αποτελεσμάτων, των επιπτώσεων της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε την έκκληση που γίνεται να συνεχίσει η δουλειά αυτή και να υπογραμμίσουμε περισσότερο τη σύνδεση ανάμεσα στις επενδύσεις και την ε, οικοδόμηση θεσμών. Αυτού του είδους οι εκθέσεις δείχνουν ότι εμείς που είμαστε Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών μπορούμε να μπούμε περισσότερο σε λεπτομέρειες όσον αφορά τα αποτελέσματα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενικά μιλώντας, αυτό είναι το έγγραφο εργασίας που εγώ σας υποβάλλω σχετικά με την ειδική έκθεση του Λεκτικού Συνεδρίου για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον εκπρόσωπο του Λεκτικού Συνεδρίου, στον κύριο Εγκβίλντα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, σας είμαι ευγνώμων κύριε Όλμπριχτ, κύριε Σιγητά, για αυτά που είπατε. Νομίζω ότι συνοψίζετε πάρα πολύ καλά την έκθεσή μας. Επίσης, είμαι ευγνώμων και για το έγγραφο εργασίας του, το οποίο νομίζω ότι ευθυγραμμίζεται απόλυτα στη δικιά μας ειδική έκθεση. Συνοψίζω τα συμπεράσματά μας σε τρία-τέσσερα σημεία. Πρώτον, συμφωνώ με τον κύριο Όλμπριχτ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει πάει αρκετά καλά δεδομένου του πλαισίου και των πολιτικών και οργανωτικών δυσκολιών που έχει να αντιμετωπίσει στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, το δεύτερο που είπε και ο κύριος Όλμπερτ είναι ότι τα προγράμματα επενδύσεων είχαν μεγαλύτερη επιτυχία από ότι τα προγράμματα οικοδόμησης ε, θεσμών στις χώρες αυτές. Καλό είναι λοιπόν στο μέλλον τα μελλοντικά επενδυτικά προγράμματα να συνδεθούν περισσότερο με το δεύτερο σκέλος, δηλαδή την οικοδόμηση θεσμών. Ένα άλλο θέμα είναι βέβαια η βιωσιμότητα των προγραμμάτων. Αυτό όμω έχει να κάνει και με τους δικαιούχου. στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθει κανείς δικό του το πρόγραμμα για να πετύχει αυτό, τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτός αυτής. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή η διοίκηση στις λόγω χώρες έχει πολλές αδυναμίες, γι' αυτό και δεν ήταν δυνατόν οι ίδιοι να προτείνουν προγράμματα. Τα περισσότερα τα προτείνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν τα νιώθω και σαν δικά τους. Και ίσως γι' αυτό να είναι και αδύναμα τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Ένα τρίτο πάντως των επιδετικών προγραμμάτων που μελετήσαμε δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν και από την άλλη κατηγορία της οικοδόμησης θεσμών εδώ θα λέγαμε ότι δύσκολα θα προχωρήσει κάποιο από αυτά. Γι' αυτό και κάνουμε συστάσεις. Συστάσεις που αντικατοπτρίζονται πάρα πολύ καλά και στην έκθεση Όλμπριτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Πιέρ Μιρέλ έχει το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Όλμπριτ πρώτα απ' όλα για την έκθεσή του. Όπως επίσης και το λεκτικό συνέδριο. Τους ευχαριστώ που επέλεξαν αυτό το θέμα πρώτα απ' όλα, το οποίο εμείς θεωρούμε σαν ένα από τα πιο σημαντικά, θα έλεγα, πολιτικό ζήτημα. Χαιρόμαστε για την αξιολόγηση του ελεγκτικού συνεδρίου, τα συμπεράσματα, τα δεχόμαστε. Όπως επίσης και τις συστάσεις που εκφράζει ο εισηγητής. Για τις πιο ειδικέ παρατηρήσεις, εφόσον μου επιτρέπετε πρόεδρε, θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά τη σύνδεση ανάμεσα στην οικοδόμηση θεσμών και τις επενδύσεις. Για μας αυτό είναι κάτι που το κάνουμε πάντα. Δεν συμφωνώ. Όταν έχει κανείς έναν ετήσιο προπολογισμό είναι δύσκολο. Και όταν τα προγράμματα οικοδόμησης θεσμών την περισσότερη φορά γίνονται σε σύνδεση με την κρατική διοίκηση, ε, κρατάνε περισσότερο καιρό οι διαδικασίες από ό,τι για τι επενδύσει. Οπότε είναι και θέμα χρόνου συχνά. Γι' αυτό και τώρα έχουμε μια πιο οτομιακή προσέγγιση, προκειμένου να συμπεριλάβουμε κάθε είδους πρόγραμμα αρρωγής, να περιλαμβάνει και τα δύο. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει. Όμως η κύρια παρατήρηση πιστεύω που περιλαμβάνεται στην έκθεση Όλβερτ αλλά και σε εκείνη του λεκτικού συνεδρίου είναι το θέμα της βιωσιμότητα. Το κύριο ζήτημα εδώ, συμφωνούμε, είναι η δυσκολία εμπλοκής των δικαιούχων. Πώς να νιώσουν δηλαδή ότι τα προγράμματα αυτά είναι δικά τους και πώς να δείξουν βούληση γι' αυτά. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για τις χώρες πραγματικά είναι δύσκολο να γίνουν μεταρρυθμίσεις σε αυτούς τους τομείς, για λόγους βέβαια που δεν θα ήθελα τώρα να σας εξηγήσω γιατί θα μας έπαιρνε πάρα πολύ καιρό. Μερικές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις πονάνε τις κυβερνήσεις των χωρών. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η δέσμευση που αναλαμβάνει η κυβέρνηση στην κάθε χώρα τηρείται κιόλα. Υπάρχει διάλογος βέβαια στη διαδικασία σταθεροποίησης προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεσμεύσει αυτές των χωρών τηρούνται. Άπαξ και υπάρχει πολιτική δήλωση, όπως για, βούληση, όπως για παράδειγμα για το θέμα των θεωρήσεων, όταν υπάρχει ένα σαφής στόχος, τότε τα προγράμματα εφαρμόζονται έγκαιρα, γιατί η ενδιαφερόμενη χώρα προσφέρει και αυτή τη δικιά της βοήθεια. Είναι αλήθεια όσα λέει η έκθεση, ότι η πολιτική βούληση είναι και το στοιχείο κλειδί. Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το κατά πόσο κάποια μέρη χώρες αυτές θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Διακοινοβουλευτική Επιτροπή με τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να φροντίσουμε το μήνυμα αυτό να περάσει στα μέλη των ε, κοινοβουλίων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και κάτι άλλο όσον αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές. Οι συστήσεις του λεκτικού συνεδρίου είναι πολύ συγκεκριμένες και ρεαλιστικές ιδίω προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι άδειε οικοδόμηση ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται δίνονται έγκαιρα. Θα φροντίσουμε να συνδεθεί αυτό με τα όσα αναφέρονται στο πρόγραμμα από την αρχή. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, συμφωνούμε απόλυτα με τα συμπεράσματα του Λεκτικού Συνεδρίου και τον εισηγητή. Για το συντονισμό των δωρητών τώρα, μεταξύ δωρητών. Μερικές φορές η Κομισιόν είναι πιο διάφανη από ό,τι τα κράτη-μέλη. Δημερός οι δωρητές εμφανίζονται τελευταία στιγμή και λένε «Α, και εμείς είμαστε εδώ και έχουμε συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουμε αυτό ή εκείνο ή το άλλο». Πολλές φορές αυτό γίνεται πολύ αργά στη διαδικασία και δεν μας βοηθάει για να έχουμε ένα καλό συντονισμό. Όμως, όντως, κάνουμε προσπάθειε σε αυτό το τομέα. Πριν από δύο εβδομάδε είχαμε μια συνάντηση με όλου του δωρητέ, έτσι ώστε να φροντίσουμε να συνεργαζόμαστε πιο στενά μεταξύ μα μέσω των αντιπροσωπιών μα επιτόπου πρώτα απ' όλα που είναι υπεύθυνε και για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Και τελευταία παρατήρηση για το θέμα της προβολής της ε, οικονομικής βοήθειας. Και το ελεγκτικό συνέδριο και ο εισηγητής δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό. Και εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία. Γιατί δεν είναι καλό μόνο να χρηματοδοτεί κανεί προγράμματα, καλό είναι να φαίνεται κιόλα, να το ξέρουν οι πολίτες στην εν χώρα τι γίνεται. Είναι πιο εύκολο να προβάλλουμε τα επενδυτικά προγράμματα παρά ε, την οικοδόμηση θεσμών. Μόνο ότι κάνουν οι αντιπροσωπείες επιτόπου με συνεντεύξει τύπου, όταν ξεκινά ένα πρόγραμμα, με ανακοινοθέντα τύπου, σε διάφορα στάδια του προγράμματος, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και ευχαρίστως να συζητήσουμε παρετέρω ό,τι βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν για να ενισχυθεί η προβολή του έργου μας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο τότε καλό βράδυ και αύριο στις 9 το πρωί θα τα ξαναπούμε.